La Commissione Petizione. Non hanno chiesto? Sì, hanno chiesto e l'ho perso. L'ho perso? Sì. Buongiorno a tutti. Diamo inizio. Καλημέρα σε όλους. Ας ξεκινήσουμε τις εργασίες της Επιτροπής, μιας και όλοι οι συνάδελφοι έχουν έρθει. Ας ξεκινήσουμε από το σημείο 8. Διαχείριση της δαπάνης που έχει να κάνει με την διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και φετέρου την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. Δίνω τον λόγο στην Ανιέσε Λεμπόν σε λίγο. Θα περάσουμε μάλλον στην ψηφοφορία της έκθεσης. 2014-2020. Πρόκειται για ένα ντοσχέ που περιλαμβάνεται στο πακέτο της υγείας ζώων και φυτών. Δεδομένου ότι η πρόταση θα τεθεί σε ισχύ τον την 1η Ιανουαρίου 2014, θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις πριν από το υπόλοιπο πακέτο. 17 τροπολογίες, 117 τροπολογίες, ε, τέσσερα πακέτα. Κυρία Ανιές, θέλετε το λόγο. συντομία κύριε Πρόεδρε, τα ουσιώδητα είπατε. Το βασικό είναι ότι ψηφίζουμε με πολύ στενό διάγραμμα αλλά τα καταφέραμε και το έργο τελικά που καταφέραμε είναι μια πολύ καλή συμβαστική λύση και Ευχαριστώ θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτό. Τη γραμματεία, την αίμα, τον Πάολο κτλ. Ελπίζω όλοι να έμειναν ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ Άγνες. Ξεκινούμε λοιπόν με τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Τροπολογίο 4. Παβόρε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Του εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία του Επιτροπής Περιβάλλοντος 5. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να το ελέγξουμε. Ξεκινώ την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 5 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 60 Πόλσον. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα πρέπει να περάσουμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 64 του Πόλσεν. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Για μία ψήφο. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 61 Κέρστιγκερ. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε το μπλοκ, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο μπλοκ, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την έξι της εισηγήτριας υπέρ με ανάταση της χειρός. Κατά, Αποχές εγκρίνεται. Όχι. Εντάξει, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει. Τροπολογία 6 της εισηγητής υπέρ. Κατά. Ναι, ναι. Απορρίπτεται. Ναι, είχες δίκιο. Ζωζέ. Περνούμε τώρα στο μπλοκ 2, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχι, άρχεται η ψηφοφορία. Δεύτερο μπλοκ, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 7. Διανατάσεως της χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 69 υπέρ της 69 της εισηγήτριας. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την budget 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τον συμβιβασμό 1. Unblock. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνούμε το μπλοκ 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 75. Γκαρσία Πέρες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπλοκ 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνούμε στην 12 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και η 12 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έμβη 13. Υπέρ, κατά, αποχές, δεν φαίνεται το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία για τη 13 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ναι, ναι κατά, μια πλειοψηφία κατά. Πέρα της ψηφοφορίας, ναι, ναι, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 14 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ, διανατάσεως της χειρός, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνούμε μετά τη 14 στη 16 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Μπαράτσου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνούμε μετά στην 15 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω. 18 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απορρίπτεται, με συγχωρείτε. Ψηφίζουμε τώρα την 83. Γκαρσία Πέρες υπέρ, κατά. Δεν φαίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 83. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 83. Τροπολογία 83. Απορρίπτεται. Ελίζαμπεθ. Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση. Η 17 ε, απορριφθηκε Ενβι NV18 απορρίφθηκε. Μήπως θα πρέπει να ψηφίσουμε τις τροπολογίες αυτές εφόσον η άλλη δεν, ε, δεν εγκρίθηκε. Ευχαριστώ Ελίζαμπεθ. Έχεις δίκιο. Πρέπει να ψηφίσουμε μετά από τη 18 Ποιοι είναι υπέρ της 18 της εισηγήτριας. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια, η 83 Γκαρσία Πέρες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Στη συνέχεια, 20 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την 84 Αγιούσο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα 86 της εισηγήτριας. 86 υπέρ. Όχι. Με συγχωρείτε, όχι. Καταπίπτει αυτή. 21 της, 22 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια, 87 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. «24 περιβάλλοντος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 περιβάλλοντος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 88 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 περιβάλλοντος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Η 26 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ναι, πολύ κοντινή. Για μία ψήφο απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 24 διανατάσεως της χειρός της εισηγήτριας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Την 90, Γκέρλινγκ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνούμε στην τροπολογία 96, Γκαρσία Πέρες και άλλοι. Υπέρ, κα, υπέρ, Α, 95 κατέπεσε. 96 Γκαρσία Πέρες υπέρ. Διανατάσεως της χειρός. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται θα έλεγα εγώ. Να ελέγξουμε. Η εισηγήτρια θέλει να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 96. Περ... Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Α, καλά έκανες, πράγματι, παρατρίχα, πέρασε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιγνάσιο. Τώρα, 99, 29, ε, με συγχωρείτε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Τροπολογία 30 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, θα έλεγα ότι απορρίφθηκε αυτή τη φορά. Την 99. Γκέρλινγκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100. Γιάρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά θα κάνουμε έλεγχο. Ελέγχουμε. Τροπολογία 100. Γιάρ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Τροπολογία 100, λοιπόν, εγκρίνεται. Περνούμε την τροπολογία 31. Η συγγήτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 101 Γκαρσία Πέρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 της εισηγήτριας υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε της Επιτροπής Περιβάλλοντος την 32, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Την 33 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. 33. Αρχίζει η ψηφοφορία. Επιτροπή Περιβάλλοντος. Α, ναι, δεν περνάει. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 103. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε. 34 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 105. Γκαρσία Πέρες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 107. Γκέρλινγκ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34. Όχι, κατέπεσε. 40. 40 της εισηγήτριας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συνεχίζουμε, 108, γκέρλινγκ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την 110, Πόλσαν, υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 110. Πόλσον. Απορρίπτεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μετά την 110 περνάμε στην 111 της εισηγήτριας. Διανατάσσεως της χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στη συνέχεια 41, 41 εισηγήτριας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 Γκαρσία Πέρες, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και στη συνέχεια περνάμε στην 43 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 Σιεκυρισκή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Την 45 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 46 επιτροπής, τη 47 της Επιτροπής Περιβάλλοντος κατά αποχές απορρίπτεται. 48 περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 116 γιάρ υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 116 γιάρ πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Ισοψηφία. 46 του εισηγητή, της εισηγήτριας, διανατάσεως της χειρός. 46. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνούμε στα παραρτήματα τώρα. Μία της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 52 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 Γκάρλινγκ υπέρ. Μια στιγμή να ελέγξουμε για την 55. Καταπίπτει 55. 56 Νταντζίλα. Υπέρ. Διανατάσσεω τη χειρός. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Την 57 Ντάντζιλα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την 57. Αρχίζει η ψηφοφορία. 57. Πέρα της ψηφοφορίας. Πολύ. Απορρίπτεται για δύο ψήφους. Τελειώσαμε. Συνάδελφοι, τελειώσαμε, αλλά μας ξέφυγε μια τροπολογία, μου λέει εδώ η γραμματεία. Πρέπει να ψηφίσουμε στη δεύτερη σελίδα, με συγχωρείτε, στην τρίτη σελίδα, τροπολογία 15 της εισηγήτριας. Μετά από την, το τρίτο μπλοκ έχουμε την 15 της εισηγήτριας. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν θα ψηφίσουμε την νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τη θέτω σε ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε τώρα το νομοθετικό ψήφισμα το οποίο μόλις ψηφίσαμε. Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την ε, έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για έγκριση σε πρώτη ανάγνωση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Ωραία. Εγκρίθηκε. Και εν τέλει ψηφίζουμε για την ε, ομάδα διαπραγμάτευσης ε, και τους σκιώδεις εισηγητές. Αρχίζει η ψηφοφορία για την ομάδα διαπραγμάτευσης. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στη συνάδελφο Λεμπρούν. Καλή τύχη στις διαπραγματεύσεις Μέχρι την 1η Ιανουαρίου πρέπει να τα καταφέρουμε. Συγχαρητήρια. Συνάδελφοι, τώρα ας περάσουμε στην έκθεση Eric Andrew. Όπως ξέρετε η έκθεση αυτή ε, περιφερειακό σήμα ποιότητας προς καλύτερες πρακτικές στις αγροτικές οικονομίες. Θα δούμε τις τροπολογίες. Ευχόμαστε μέχρι την ε, συνεδρίαση των συντονιστών στις 5 Δεκεμβρίου να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβάλαμε για την τροπολογία του ονόματος της ονομασίας για, να, για τη διαγραφή του όρου ποιότητας. Έτσι αποφασίσαμε στην συνεδρίαση των συντονιστών και ζητήσαμε να λέγεται περιφερειακό σήμα, όχι περιφερειακό σήμα ποιότητας. Έρικ, θα πάρεις το λόγο. Ναι. Ένα λεπτό. Oui, merci, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, κυρίως τους χειώδεις ηγητές, για την ε, συνεργασία τους, γιατί έτσι καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις αρχικές παρεξηγήσεις μας. Και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Γραμματεία για την ε, ανεκτήμητη συμβολή της καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ, Ερικ. Αν είσαστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ας ξεκινήσουμε από, τον, από τους συμβιβασμούς. Όχι? Όχι, όχι, από την παράγραφο 1, συγγνώμη. Τροπολογία 44, Ρένες, Ρέιμερς, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 47, Ρέιμερς, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 48. Γκάμπριελ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σε μπλοκ τώρα. Ε, συμβιβαστική τροπολογία. Για την παράγραφο 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνούμε στην τροπολογία 53. Σεντό ή Άλαμπαρτ. Ποιοι είναι υπέρ. Διανατάσσεως της χειρός. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνούμε στη, συμβιβαστική πρόταση για την παράγραφο 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 63, Ντάντσιλα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 63. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ah, oui. ne passe pas. Okay. Έχεις δίκιο, ε. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται η τροπολογία 63. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 65 Αντριού. Διανατάσσεως της χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το συμβιβαστική πρόταση για την παράγραφο 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνούμε στην τροπολογία 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 Νταντσίλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική πρόταση για την παράγραφο 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 76 σκοτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 86 σκοτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σε μπλοκ τώρα συμβιβαστικές προτάσεις για την παράγραφο 7 και το 7α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 98 Μπαράτσου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 99 Νταντζίλα υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται, ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 100 Σκοτά υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ρέιμερς υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Reimers υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Τζόχανσον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Νταντά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Πατράου Νέβες υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Αντριού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Νταντζίλα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Γιώχανσον υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 13 του Γιώχανσον. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε για μία ψήφο. Τροπολογία 14 Ρέιμερς υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για τη 14. Ναι, αρχίζει η ψηφοφορία για τη 14. Πρέπει να είναι πολύ κοντά, ναι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Είχαμε δει καλά. Ε, τροπολογία 15. Χέραντς Καρσία και άλλων. Υπέρ. Διανατάσεως. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ρέιμερς. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Πατράου Νέβες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Γέγκλε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Σκοτά υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Νίκολσον υπέρ, κατά θα έλεγα πως εγκρίθηκε. Τροπολογία 21. Σκοτά. Υπέρ. Κατά. Hm. Έλεγχος για την 21 σκοτά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Όχι, όχι. Απορρίπτεται. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όμως. Απορρίφθηκε, εντάξει. Τροπολογία 22 ε, Νίκολσον υπέρ διανατάσεως κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 Έρανς Γκαρσία και άλλον. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 Ρέιμερς υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Δεν είμαι σίγουρος. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 23 Reimers. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Πατράουν υπέρ, διανατάσεως κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Γκουλάγα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το συμβιβασμό για την αιτιολογική σκέψη H. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 32 Ντάντζιλα, ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 42 Γκουλάγ, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 38, Νταντά, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40, Χάουσλινγκ Μποβέ, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 40. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 40. Η Αντιπρόεδρος εδώ ψήφισε τον, ε, καταψήφισε τον εαυτό της. 40 ε, αρχίζει ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Αρνητικό το αποτέλεσμα για μία ψήφο. Τροπολογία 41 Γκάμπριελ υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. 43 Μπαράτσου υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την ε, Ρέτζι τη γνωμοδότηση. Θα... Ναι, ναι, είναι ξεχωριστές οι ψηφοφορίες. Ρέτζι, η πρώτη. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε τη Ρέτζι 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 5. Υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται και αυτή. Ρέτζι 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Και 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Περνούμε στην... Ποια? Ωραία. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη Ρέτζι 9. Αρχίζει η ψηφοφορία. Περατούται η ψηφοφορία. Μπράβο σας, εγκρίθηκε. Η 9 εγκρίθηκε. Είσαστε προσεκτικοί. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Ας ξεκινήσουμε. Τραν γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τράνα 1 και 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τράν 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τραν 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 8 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω. Έλεγχος. Έλεγχος για την τραν 8. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για να δούμε. Πέρα της ψηφοφορίας, εγώ θα λέγα πως απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. Και τέλος, τραν 10, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε υπέρ ηλεκτρονικά. Με συγχωρείτε, ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ομόφωνα. Όχι. Τρεις ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια, Έρικ. Μπράβο σου. Φυσικά αναμένουμε και την απόφαση στις 5 Δεκεμβρίου και ελπίζω ότι οι πρόεδροι των ομάδων δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα με την αλλαγή του τίτλου. Φτάνουμε τώρα στο σημείο 10, ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Ο κύριο Τάσο Στανιώτη, είναι μαζί μας. Καλημέρα. υπάρχει η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πολλοί από εμά την περασμένη εβδομάδα εξέφρασαν την αμηχανία τους μπροστά στα σχέδια των ε, πράξεων ε, εξουσιοδότηση της Επιτροπής και έτσι ζητήθηκε αυτή η ανταλλαγή απόψεων την περασμένη εβδομάδα υπήρξε μια μεγάλη πλειοψηφία κρατών μελών ε, στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας ε, που εξέφρασαν κάποιες ε, αντιρρήσεις για το κατά πόσο συμφωνούν οι πράξεις κατεξουσιοδότηση με το θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Τάσο Χανιώτη, για να μας δώσει επεξηγήσεις για, για το σημείο που βρίσκονται οι σχετικές ε, συνομιλίες, για τις αντιρρήσεις, για τις δυνατότητες τροποποίησης πριν από την επίσημη υιοθέτηση των κατεξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή και τη διαβίβασή τους στο Κοινοβούλιο. Ήδη από τώρα συνάδελφοι σας ανακοινώνω, προσοχή προσοχή, ότι αυτή η πρώτη ενημερωτική συζήτηση θα οδηγήσει σε ακόμα πιο αναλυτική συζήτηση στις 2 Δεκεμβρίου. Σήμερα απλώς ενημερωτικά συναντιόμαστε. Ο Διευθυντής κύριος Τάσος Χανιώτης θα μας ενημερώσει. Στις 2 όμως Δεκεμβρίου θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη το θέμα ε, ε, μια συζήτηση μάλλον με την Επιτροπή και με τις υπηρεσίες γεωργίας και κλεισμένων των θυρών για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Θα μπορέσουμε να κάνουμε ε, παρατηρήσεις επί της ουσίας για να επηρεάσουμε τη διατύπωση των πράξεων αυτών. Αν και υπενθυμίζω, όταν οριστικοποιούνται και υιοθετούνται επίσημα από την Επιτροπή η κατεξουσιοδότηση πράξης, το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα ή να τις υιοθετήσει ή να τις απορρίψει, όχι να τις, μετα... να τις τροποποιήσει. Ε, μεταξύ άλλων, συνάδελφοι, στη συνάντηση των συντονιστών θα συζητήσουμε και με τον Επίτροπο Τσόλος στις 9 Δεκεμβρίου. Ε, ο λόγος πάει στον κύριο Τάσο Χανιώτη, λοιπόν. Επαναλαμβάνω γιατί βλέπω μία αμηχανία στο κρατήριο. Ενημερωτική συζήτηση σήμερα με τον κύριο Τάσο Χανιώτη την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου συζήτηση και κλειμένων των θυρών με, την, το επιτελείο του Επιτρόπου Τσόλος με εμπειρογνώμονες και άλλους εκπροσώπους της DG Agri. Στις 9 Δεκεμβρίου στη συνάντηση των συντονιστών με τον Επίτροπο Τσόλος θα ξανασυζητηθεί το θέμα. Κύριε Χανιώτη, έχετε το λόγο. Thank you, Chairman. Uh, and thank... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που οριοθετήσατε και το πλαίσιο της δικής μου παρέμβασης. Θα είμαι λακωνικός. Θα περιοριστώ σε τρία σημεία. Καταρχήν, ακούσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τα επιχειρήματα που εκφράσατε την περασμένη εβδομάδα και τις ανησυχίες σας για να φροντίσουμε έτσι να διευκρινίσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τρία επιμέρους σημεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα μαζί σας ότι στόχος των κατεξουσιοδότηση πράξεων δεν είναι να αντικαταστήσουν διατάξεις της βασικής πράξης, αλλά να τις συγκεκριμενοποιήσουν αυτές τις διατάξεις όπου δει. Οπότε και το γράμμα των βασικών πράξεων, αλλά και το, από το πνεύμα των διαπραγματεύσεων ε, δεσμεύουν όλα τα κοινωτικά θεσμικά όργανα και φυσικά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το ιδεώδες μέρος και η ιδεώδες ευκαιρία ε, να συγκεκριμενοποιήσουμε κάποια θέματα είναι η κατεξουσιοδότηση πράξη. Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για τη βασική ε, πράξη και την λογική της. Και έτσι γίνεται κυρίως στην ε, ομάδα εμπειρογνωμών. Εκεί εξετάζονται οι κατεξουσιοδότηση πράξη σε πολύ πρόωρα στάδια της εκπόνησής τους. Και μάλιστα σήμερα έχουμε μια νέα συνεδρία εμπειρογνωμόνων για τις άμεσες πληρωμές που γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και εξετάζουν το αναθεωρημένο κείμενο. Το κείμενο αυτό θα υποστεί δεχομένως και νέες τροπολογίες αν το απαιτήσει αυτό η έκβαση των συζητήσεων στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Και σε αυτές ακριβώς τις ομάδες εμπειρογνωμόνων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευκαιρία να εξηγήσει την λογική των ε, άρθρων που προτείνει. Τα κράτη-μέλη και εκπρόσωποι Ευρωπαϊ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προσωπείται πλήρως ως κανονικό, τακτικό μέλος των ομάδων εμπειρογνωμών και όχι ως παρατηρητής απλώς, έχουν την ευκαιρία λοιπόν όλοι να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, τις διαφωνίες τους, τον προβληματισμό τους. Και από όλη αυτή τη διαδικασία μπορούμε από κοινού να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που θα είναι αποδεκτό από όλους. Τέλος, θα ήθελα ευκαιρία να επιθυμίσω αυτό που είπε ο Επίτροπος Τσόλος στην Ολομέλεια της ε, περασμένης εβδομάδας και τόνισε και ο Πρόεδρος πριν από λίγο. Θα συνεχιστεί η ενημέρωση, θα έχουμε νέα ενημερωτική συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να σας ε, δώσουμε πολύ περισσότερες ε, διευκρινείς και λεπτομεριακές εξηγήσεις για την πορεία των συζητήσεων. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ τους συναδέλφους και ευχαριστώ τον Τάσο για τις διευκρινήσεις αυτές. Στις 2 Δεκεμβρίου και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση όπου θα συζητήσουμε επί της ουσίας με το επιτελείο του Επιτρόπου και με την DG Agri, τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Στη συνέχεια, για άλλη μια φορά στις 9 Δεκεμβρίου, κατά τη συνάντηση των ε, συντονιστών με τον ίδιο τον Επίτριο μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Θέλει να παρέμβει κάποιος. Σας θυμίζω ότι η συζήτηση επί της ουσίας θα γίνει τη Δευτέρα. Βέντες και George Λάιον, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο περιεχόμενο. Απλά θα ήθελα να πω ότι το πολιτικό κείμενο, η πολιτική συμφωνία θα πρέπει να τηρείται και δεν θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να γίνει ερμηνεία ε, διαφορετική στην ε, μεταρρύθμιση της ε, Γεωργίας, γιατί εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Θα πρέπει η Κομισιόν να γνωρίζει ότι από τη συνθήκη έχουμε το δικαίωμα να αποσύρουμε πράξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αλμπέρτ. George Lyon και στη συνέχεια την Νίκολσον. Ε, ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Τάσο. Ε, δεν θα αναγνωρίζει στο γεγονός ότι 18 κράτη-μέλη υπέγραψαν την ε, κοινή ε, διακήρυξη ε, όπου αναφέρουν τις ανησυχίες τους ότι η Κομισιόν κατά την έκδοση κατευθυνότηση πράξεων ξεπερνάει τα όρια της πολιτικής συμφωνίας όπως την ερμήνευαν αυτοί. Μήπως μπορείς να σχολιάσεις γιατί τα κράτη-μέλη έπρεπε να κάνουν κάτι τέτοιο. Μήπως μπορείς να μας εξηγήσεις εάν ε, έχετε ασχοληθεί με τις ανησυχίες αυτές. Διότι για 18 κράτη-μέλη υπάρχει σημαντική ανησυχία σχετικά με την κατεύθυνση ε, που παίρνει η Κομισιόν. Ευχαριστώ, George, Jim Nicholson και στην συνέχεια Κάπουλας και εδώ παρακείμενος. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι θα συζητήσουμε επί της την επόμενη εβδομάδα, οπότε δεν έχει νόημα να επαναλαμβανόμαστε. Εάν η Κομισιόν πιστεύει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τότε με εκπλήσει η θέση που παίρνει. Και μπορεί να μην είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε αυτό. Ίσως να πρέπει να συζητήσουμε αργότερα ποια είναι η θέση μας όσον αφορά τις κατεξιοδότηση πράξης. Εάν στι εκτελεστικέ πράξει έχουμε απλά καθεστώ παρατηρητή, δεν θα πρέπει στι κατεξοδότηση πράξη να έχουμε κάτι παραπάνω. και με όλο το σεβασμό προς την Επιτροπή προσπαθώ να το πω διπλωματικά. Το να έρχεται η Επιτροπή εδώ και να μας λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τη στιγμή που 18 κράτη-μέλη ε, με την υποστήριξη άλλων δύο κρατών μελών ε, έχουν ε, υπογράψει διακήρυξη όπου εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την ερμηνεία από τον Επίτροπο της Πολιτικής Συμφωνίας που έγινε τον Ιούνιο. Όλοι γνωρίζουμε, όλοι όσοι είμαστε εδώ, ξέρουμε ότι ήταν μια πολύ ευαίσθητη συμφωνία, οποιαδήποτε στρέβλωσή της, σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο ε, να την ε, δεχτούμε η Κομισιόν ε, λοιπόν ε, δεν ε, θα πρέπει να έρθει εδώ και να προσποιείται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τη στιγμή που όλοι οι άλλοι συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ, Τζιμ. σε κατανοώ απόλυτα. Λουίς Καπούλας. Ευχαριστώ. Έχω μια, ένα γνωστό ρητό που λέει ποτέ δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για να προκαλέσει την πρώτη καλή εντύπωση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση αυτή έχασε την ε, ευκαιρία, την πρώτη ευκαιρία για την πρώτη καλή εντύπωση και δεύτερη ευκαιρία δεν έχει. Και μετά την ε, πολύ ε, επίπονη κατάληξη συμφωνία με καλή βούληση από όλες τις πλευρές, μετά τις... τον κόδωρο του κινδύνου που έχει κρουστεί μετά τις πρώτες κατεξοδότης πράξεις, ε, αντιδράσαμε ομόφωνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια. Βέβαια, εκτιμώ ιδιαίτερος, εκτίμησε ιδιαίτερος αυτά που είπε ο Επίτροπος Σόλος στο Στρασβούργο και Επίσης ε, αυτά που επιβεβαίωσε με τις δικές του δηλώσεις ο κύριος Χανιώτης. Ελπίζω να είναι αυτή η γνήσια θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μην είναι απλώς η αντίδραση της Επιτροπής στην αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω τελικά να βρούμε μια ευκαιρία για να, να εκμεταλλευτούμε έστω και μια δεύτερη ευκαιρία για να αναμορφώσουμε την πρώτη κακή εντύπωση. Ευχαριστώ Λουίς. Πραγματικά η φράση σου ήταν πολύ εύστοχη. Κύριε Σεκέρσκι. Θα ήθελα να ρωτήσω για αυτή την ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Γιατί ομολόγω την ε, άγνοιά μου εδώ. Ποια είναι η σύνθεση αυτής της ομάδας εμπειρογνωμόνων και ποιος συγκαλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Και είναι η ίδια ομάδα εμπειρογνωμόνων ή διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο. Γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είναι διαφορετικοί οι εμπειρογνώμονε για κάθε θέμα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, η σύνθεση τη ομάδα εμπειρογνωμόνων και ποιο τη συγκαλεί. Δεύτερον, τι γίνεται με την προσέγγιση ε, των κατεξουσιοδότη πράξεων για άλλου τομεί, ε, για την Επιτροπή περιφερειακή ανάπτυξη, την Επιτροπή Μεταφορών, α πούμε. Εκεί η προσέγγιση άλλων επιτροπών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα των κατά εξουσιοδότηση πράξεων επίσης ε, είναι, ε, δημιουργεί ερωτηματικά και ανησυχίες. Γιατί εμείς είχαμε μεγάλο προβληματισμό. Συμμερίζονται αυτές τις ανησυχίες και άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τις κατά εξουσιοδότηση πράξεις. Ο κύριος Μπλάτενφέλντερ και μετά ο κύριος Άγνιο και είναι ο τελευταίος μας ομιλητής. Nem csupán a közös agrárpolitika szempontjából aggályos, hanem aggályos az unió όχι μόνο από την πλευρά της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής είναι ανησυχητική η ερμηνεία αυτά, αλλά ε, έχει να κάνει και με την όλη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η Κομισιόν ε, έχει ανατρέψει την λεπτή ισορροπία που βρέθηκε. Έτσι λοιπόν... Ε, δημιούργησε ένα στρατόπεδο ε, ανθρώπων που είναι ε, σκεπτικοί απέναντι στην Κομισιόν, πέρα από τους ευρωσκεπτικιστές που έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν συνέπειες, διότι ε, ταράχτηκε η πολιτική εμπιστοσύνη και δεν θα είναι εύκολο να αποκατασταθεί. Θα, πρέπει να κάνει λοιπόν πολύ περισσότερα η Κομισιόν για να φροντίσει να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Αγνιέ. Πρόεδρε, ε, υποστηρίζω όλα τα μέλη, τα μέλη που έχουν ήδη λάβει τον λόγο. Ασυνήθιστο για μένα, θα σας ξεχνιάσει αυτό. Αυτό που με ανησυχεί εδώ είναι αυτή η τεράστια γραφειοκρατία που ονομάζεται Επιτροπή ελέγχει ε, πώς έχει το τοπίο ε, κάθε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί κάθε φορά έρχεται και ταράζει τα νερά. Ευχαριστώ. πάλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση. Σύμφωνα με τις ε, δικές μου πληροφορίες, 23 κράτη-μέλη έχουν εκφραστεί επικριτικά. Ίσως ε, τα τελευταία πέντε να μην έχουν ασχοληθεί ακόμα με το θέμα αυτό. Ε, προς τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, θα ήθελα να θέσω την εξής ερώτηση. Ε, βρήκα θετικό ε, το ότι θα πρέπει να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στις κατεξοδότηση πράξης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που το Κοινοβούλιο έχει μόνο καθεστώς ε, παρατηρητή. Ε, αυτό δεν ε, είναι ακριβώς ενεργός συμμετοχή. Και το τελευταίο καιρό έγινε γνωστή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η αντίσταση των κρατών μελών και αυτό είναι κάτι το οποίο συμφέρει τους ευρωσκεπτικιστές. Η Επιτροπή λοιπόν ε, θα φροντίσει να συμμετέχει στις δημοκρατικές εξελίξεις ε, στην Ευρώπη. Πού, γι' αυτό, γι αυτό λέει είναι και η Κεντρική Επιτροπή. Ευχαριστώ, Μία ερώτηση έχω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφόσον όλοι μιλούν τόσο πολύ, το έχουμε συζητήσει και κεκλεισμένων των θυρών, θα ήθελα να ξέρω τι πρόβλημα έχει η Επιτροπή. Γιατί δεν μπορούμε να επανέλθουμε στα όσα συμφωνήσαμε. Ποια είναι η βάση εδώ. Γιατί πρέπει να τα αλλάξετε όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ρουμπίξ, ο Μάρτιν äh, Ναι. Ε, και εγώ βρίσκω η υπερβολική την ε, σύγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με μια κεντρική ε, επιτροπή απολυταρχικού κράτους. Ίσως ε, θα μπορούσε ο εκπρόσωπος Επιτροπής ε, να μας κάνει κάποια διευκρίνηση. Ε, είπε ότι θα συμμετέχουμε ενεργά. Όχι, παρατηρητές θα είμαστε. Εάν ως Κοινοβούλιο συμμετέχουμε ενεργά, αυτό όντως θα δείξει την καλή βούληση. Νομίζω ότι εδώ μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Θα ξαναδώσω το λόγο φυσικά στον Διευθυντή Τάσο Χανιώτη. Θα ήθελα ωστόσο να πω και εγώ μερικά πράγματα. Καταρχήν ε, πάνω στο επιχείρημα αυτό εκ μέρους όλων μας υπάρχει ε, απόλυτη σύγκληση απόψεων. Ε, όπως φάνηκε και από όλους τους παρεμβαίνοντες υπάρχει μια βούληση ξεκάθαρη να, να, εξασφαλίσουμε ότι η κατεξουσιοδότηση πράξης ε, δεν είναι πολιτικές πράξεις, ε, είναι εφαρμοστικές διατάξεις ε, πολιτικών αποφάσεων. Αυτό είναι θεμελιώδος και θα το επαναλάβουμε και στην έκθεση Ζάιερ σε λίγες εβδομάδες. Συνάδελφοι, ας μην ξεχάσουμε ότι, ας μην ξεχνάμε ότι οι πράξεις κατεξουσιοδότηση υπήρξαν κατάκτηση του Κοινοβουλίου μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας και εν τέλει αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι μπορούμε να τις απορρίπτουμε. Ε, δεν είναι και πια και κανένα καμιά τεράστια τραγωδία. Δεν πρόκειται για απόρριψη νομοθετικής πράξης που σημαίνει ότι ξαναξεκινούμε από το μηδέν, πρώτη ανάγνωση, δεύτερη ανάγνωση κτλ. Ε, πρέπει να ε, συνηθίσουμε ε, να έχουμε μια ηρεμία πνεύματος. Εάν απορρίψουμε μια κατεξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή μετά από λίγες εβδομάδες θα μας παρουσιάσει, θα μας υποβάλει μια άλλοι. Ε, η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε στα τέσσερα, μάλλον πέντε νομοθετικά κείμενα της κοινή γεωργικής πολιτικής, αν λάβουμε υπόψη μας και τις μεταβατικές διατάξεις, έχουμε ασχοληθεί με τεράστιο αριθμό κατεξουσιοδότηση πράξεων. Θα πρέπει λοιπόν να εκτελούμε τον ρόλο μας, αλλά να μην ανησυχούμε πια και αν είμαστε αρνητικοί απέναντι σε κάποιες πράξεις κατεξουσιοδότηση. Ε, θυμίζω, παραμένει κατάκτηση κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση στις εκτελεστικές πράξεις, όπου δεν έχουμε καμία δυνατότητα παρέμβασης εκεί. Με αυτές τις διευκρινήσεις λοιπόν ε, θα δώσω το λόγο στον Τάσο και θα του ζητήσω να απαντήσει, ε, αν και επαναλαμβάνω, επί της ε, ουσίας ίσως και η γραμματεία θα μπορέσει να μας ε, βοηθήσει συνοψίζοντας τα βασικά σημεία για να προετοιμάσουμε τη συζήτηση επί της ουσίας την Δευτέρα στις 2 Δεκεμβρίου γιατί στη συζήτηση εκείνη θα αντιμετωπίσουμε ένα προς ένα όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Τάσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, δεύτερη ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω μερικές διευκρινήσεις που φαίνεται ότι με την πρώτη μου απόπειρα δεν κατάφερα να δώσω. Ε, δεύτερη προσπάθεια λοιπόν. Καταρχήν το πρώτο πράγμα που πρέπει να, δια, να διασαφηνίσουμε είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούμε. Η βασική πράξη είναι η βασική πράξη. Τελεία και παύλα. Αυτό μας δεσμεύει όλους. Δεν συζητούμε τίποτα έναντι των ε, βασικών πράξεων. Αυτό που συζητούμε είναι κάποιοι τομείς για του οποίου χρειάζονται λεπτομέρειες που δεν βρίσκονται στη βασική πράξη. Και αυτοί οι τομεί χρήζουν διευκρινήσεως. Αυτές οι λεπτομέρειες πρέπει να αποσαφινιστούν. Και σήμερα είναι η πρώτη φορά που η ομάδα εμπειρογνωμόνων συζητά την ενοποιημένη εκδοχή το, της πρότασης ε, για την καταξιδότηση πράξης. Αυτό που συζητούμε στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις είναι επιμέρους ε, ε, άρθρα είναι συντακτική προσπάθεια. Και όταν έχουμε προτάσεις άρθρων για συζήτηση, θα πρέπει να διευκρινιστούν κάποιοι τομείς, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές σε άλλα σημεία και σήμερα έχουν γίνει προτάσεις για τροποποίηση. Και σίγουρα σε άλλους τομείς θα χρειαστούν περαιτέρω αλλαγές. Σε ορισμένα σημεία φυσικά το κείμενο θα μείνει αμετάβλητο. Και ελπίζω να καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι έχει λογική αυτό που κάνουμε. Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για απόπειρα τροποποίησης της βασικής πράξης. Κανείς δεν έχει ούτε τη βούληση, ούτε καμία πρόθεση να κάνει κάτι τέτοιο, να αλλάξει τη βασική πράξη. Είπα, ρωτήσατε προηγουμένω, αν εσεί ε, συμμετέχετε πλήρω σε αυτέ τι ομάδε. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για ομάδα εμπειρογνωμόνων. Αυτή θα συζητήσει το θέμα. Στην ομάδα εμπειρογνωμόνων συμμετέχουν εμπειρογνώμονε από τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν πληροφορίε σε όλες τις φάσεις των προτάσεων ε, για, όλες, για όλα τα σχέδια. Τις ίδιες πληροφορίες και ταυτόχρονα τις λαμβάνετε κι εσείς. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εκπρόσωποι σας στην ομάδα εμπειρογνωμόνων έχουν δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να εκφέρουν τη γνώμη τους. Εσείς αποφασίζετε ποιου θα ορίσετε εκπροσώπους σας. Όχι εμείς, αλλά μιλούμε για εμπειρογνώμονες, όχι για ευρωβουλευτές και οι εμπειρογνώμονε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν την ίδια ευκαιρία με του υπόλοιπου εμπειρογνώμονε να εκφράσουν τι ανησυχίε του αν υπάρχουν. Και έχουμε περιπτώσει που έγινε κάτι τέτοιο. Εκφράστηκαν ανησυχίε. Τώρα, ποια είναι η επόμενη φάση, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε πώ θα εξελιχθούν σήμερα οι συζητήσει για την ενοποιημένη πρόταση, ενοποιημένη εκδοχή, για ποιους τομείς χρειάζονται διευκρινήσεις ε, ή υπάρχουν ανησυχίες και θα προβλεφθεί και δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για να συνεχιστεί η, εργασία και η εξέταση του ενοποιημένου κειμένου. Ήδη έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Ήδη ε, θα γίνουν κάποιες ε, διευκρινήσεις και ελπίζω με όλα αυτά να καταλήξουμε σε μια σωστή εξήγηση. Νομίζω ότι κάλυψα τα ερωτήματά σας. Τώρα, ο George Lyon έκανε μια ερώτηση, αλλά που απευθύνεται περισσότερο στα κράτη-μέλη παρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αν δείτε τις λεπτομέρειες θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στις κατεξοδότηση πράξεις που αφορούν συγκεκριμένα κράτη-μέλη, όχι όλα τα κράτη-μέλη. Και στη συζήτηση αυτό που κάνουμε και αυτό που έχουμε την ευθύνη να κάνουμε είναι να δούμε αν οι διευκρινήσεις που δώσαμε και οι αλλαγές που κάναμε έχουν νόημα στη συζήτηση. Και επαναλαμβάνω, η διαδικασία δεν έχει διεκπαιρεωθεί, βρίσκεται να εξελίξει. Γιατί μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο και ότι έχει αποφασιστεί και ήδη είναι όριμο και ψηφοφορία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ Τάσο Χανιώτη. Θα ήθελα να διευκρινίσω ωστόσο ότι το άτομο που εκπροσωπεί το κοινοβούλιο, ο εμπειρογνώμονας, δεν έχει πολιτική εντολή και δεν έχει καμία δυνατότητα παρέμβασης. Είναι σαφές αυτό. Δεν μπορεί να παρέμβει γιατί δεν έχει εντολή, δεν έχει εξουσιοδότηση. Ε, μπορεί μόνο να ακούσει, να αναφέρει τι έγινε στο σώμα των συντονιστών και οι συντονιστές μετά μπορούν να συζητήσουν με την Επιτροπή τι θα κάνει. Δεν στέλνουμε έναν εισηγητή με μια συγκεκριμένη εντολή. Είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη έχουν ομάδες εμπειρογνώμων και προσυποκότητες ε, ε, που μπορούν πολύ πιο αποτελεσματικά να δράσουν σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Εμείς έχουμε μία γραμματεία, τον Πάολο Ρώση και κάποιους συνεργάτες, αλλά περιορισμένο αριθμό ατόμων σε σχέση με τους πόρους που διαθέτει το κράτος μέλος, τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό πρέπει να τα βρούμε. Διαφορετικά οι πράξεις κατεξουσιοδότηση της Επιτροπής θα απορρίπτονται. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα να επηρεάσουμε και έχουμε τόσα πολλά άλλα πράγματα να κάνουμε. <clears throat> Όταν έχουμε 20 ε, κράτη-μέλη που θεωρούν ότι η Επιτροπή ξεπέρασε τα όρια της αρμοδιότητάς της, της εντολής της και τα διαβάσαμε τα επιχείρηματά τους. Εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας θα μιλήσουμε τη Δευτέρα. George. Really Ε, τα έχω λίγο χαμένα τώρα με το θέμα της εκπροσώπησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή των κατεξιοδότησε πράξεων. Εγώ αρχικά πίστευα, ή ε, τουλάχιστον έτσι μου είχε πει η γραμματεία, ότι δεν έχουν δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις αυτές ε, οι δικοί μα εκπρόσωποι. Ενώ ε, και ο Τάσο επιβεβαίωσε ότι έχουν δικαίωμα λόγου. Εγώ δεν θυμάμαι οι συντονιστές να συζήτησαν ουδέποτε ότι δεν θα επιτρέψουμε στη γραμματεία μας, στου ε, εκπροσώπους μας να λάβουν το λόγο στις συνεδριάσεις αυτές. Δεν θυμάμαι να συζητήσαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να λάβουμε εμείς απόφαση αν δικαιούνται να μιλήσουν ή όχι. Γιατί αν είναι να λάβουμε τέτοια απόφαση θα πρέπει να το συζητήσουν οι συντονιστές για το αν θα έχουν δικαίωμα λόγου ή όχι εκπρόσωποι μας εκεί και τι εντολή θα έχουν να μιλήσουν. Γιατί διαφορετικά οι ανησυχίες που έχουμε δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Αν μου λέτε ότι υπάρχουν ανησυχίε ότι έχει διαταραχθεί η πολιτική συμφωνία. Μπορεί οι πυρογνώμονε μα να μην μπορούν να μιλήσουν για πολιτικά θέματα, αλλά μπορούν να πούν ε, αν ένα συγκεκριμένο θέμα ανταποκρίνεται στι ε, διαπραγματεύσει και στι θέσει των πολιτικών ομάδων. Θα πρέπει λοιπόν να αποσαφηνίσουμε ποιο ε, θα εξουσιοδοτεί στη γραμματεία μα θα λαμβάνει το λόγο στι συνεδριάσει αυτέ. Γιατί αυτά που άκουσα πριν από λίγο από τον πρόεδρο με μπέρδεψαν. Δεν ξέρω αν έχουν δικαίωμα λόγου ή όχι. Γιατί από αυτά που μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι έχουν δικαίωμα λόγου οι εκπρόσωποι μα εκεί. Θα πρέπει ίσω εμεί να του εξουσιοδοτήσουμε να μπορούν να ασκούν αυτό το δικαίωμα. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το δούμε αυτό. George. Ε. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Για να τα ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας, ο, ο, ο, της γραμματείας που συμμετέχει ως παρατηρητής δεν μπορεί να παρέμβει. Το επαναλαμβάνω, δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να παρέμβει, δεν έχει πολιτική εντολή. Και το είπα εγώ, ενημέρωσα τον Τάσο, του το λέω. Δεν μπορεί. Ε, μπορεί βέβαια άτυπα να το κάνει, αλλά δεν έχει εντολή εκπροσώπησης, δεν είναι εξουσιοδοτημένος, δεν νομιμοποιείται να μας εκπροσωπήσει. Στην έκθεση Ζάιερ θα έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον να αποφασίσουμε ως Κοινοβούλιο να ορίζουμε εισηγητές για τι κατεξουσιοδότηση πράξεις, αλλά στη διαδικασία όπως έχει σήμερα δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Αυτό που γίνεται είναι ότι ο πυρογνώμονα μα μεταφέρει τι συζητήσει και μετά κάνουμε μια πολιτική συζήτηση μεταξύ μας. Ο, εμ, ο παρατηρητής δεν είναι υπάλληλο, δεν είναι εκπρόσωπος, δεν είναι δικός μας πολιτικός υπάλληλο, είναι τυπικά συμμετέχει εκεί ως παρατηρητής και πρέπει η Επιτροπή να προσέχει πάρα πολύ να ε, ε, αναπαράγει πιστά ε, τις βασικές πράξεις στην κατεξουσιοδότηση πράξη. Γιατί διαφορετικά από τα πρώτα σχέδια των σχετικών πράξεων και τα κράτη-μέλη αλλά και εμείς είδαμε ότι δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα και εκφράσαμε τις ανησυχίες μας. Όπως Είπα, στις 2 Δεκεμβρίου θα γίνει η συζήτηση επί της ουσίας. Στις 9 Δεκεμβρίου ε, και κλεισμένων των θυρών οι τονιστές θα κάνουν μια αξιολόγηση με τον Επίτροπο και στη συνέχεια θα έχουμε κάθε δυνατότητα, όχι μόνο για να διορθώσουμε αυτές τις πρώτες στην πράξη, αλλά και για να καταστρώσουμε μια στρατηγική παρακολούθηση ελέγχου, ε, μια δική μας στρατηγική, για να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον τέτοια προβλήματα με τα πρώτα σχέδια των κατεξουσιοδότης συμπράξεων. Καλώς, Τζιμ, θέλεις και εσύ να πάρεις το λόγο, παρακαλώ. part, uh, Από ό,τι καταλαβαίνω, όλοι γνωρίζουμε που βρισκόμαστε σήμερα 26 Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Θες να λυθούμε και με τον Επίτροπο. Αλλά εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, πριν τις 13 Μαρτίου του χρόνου δεν πρόκειται να προχωρήσουμε πάνω στις κατεξοδότηση πράξεις. Εμένα έτσι μου είπαν την προηγούμενη εβδομάδα. Αν ισχύει αυτό, τότε θα έχουμε μία συνεδρίαση της Επιτροπής και μία σύνοδο στο Στρασβούργο για να ε, ασχοληθούμε με το θέμα. Αυτό εμένα δεν μου φαίνεται ότι είναι πολύς χρόνος και μάλλον θα πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό αργότερα. Μην ξεχνάμε το χρονοδιάγραμμα, διότι μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος θα έχει και πολλές άλλες δουλειές. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ευθύνες μας και τι χρονοδιάγραμμα έχουμε. Και εδώ σε ευχαριστώ Τζίμα που μου δίνεις τη δυνατότητα να διευκρινίσω την πορεία. Τον Μάρτιο θα έχουμε την έγκριση της πράξης κατά από το Συλλογικό Σώμα της Επιτροπής. Από τη στιγμή που τυπικά, επίσημα, η Επιτροπή θα υιοθετήσει, θα εγκρίνει την κατεξουσιοδότηση πράξη, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Μπορούμε μόνο να καταψηφίσουμε ή να υπερψηφίσουμε. Η δουλειά πρέπει να γίνει πριν. Πρέπει να την κάνουμε τώρα και πρέπει να την κάνουμε στην επόμενη συνάντηση. Όταν θα εξετάσουμε καινούργια κείμενα, καινούργια σχέδια κειμένων, να μπορούμε να κάνουμε τις υποδείξεις μας και τις παρατηρήσεις μας για να επηρεάσουμε την επιλογή της κατεξουσιοδότησης πράξης. Όταν φτάσουμε το Μάρτιο, τα πράγματα θα έχουν τελειώσει το τελικό κείμενο, η τελική πράξη που θα έχει υιοθετηθεί από την Επιτροπή, εάν δεν μας ικανοποιήσει, μπορούμε να το απορρίψουμε. Η δουλειά όμως που πρέπει να κάνουμε αυτές τις εβδομάδες είναι να προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε αυτά τα πρώτα σχέδια. Το είπε και ο Τάσος. Είναι τα πρώτα σχέδια, τα πρώτα κείμενα που κυκλοφορούν. Φυσικά θα έρθουν και καινούρια. Ήδη γίνεται λόγος για ένα νέο σχέδιο πριν από τα Χριστούγεννα. Θα δούμε τι θα, πώς θα είναι γραμμένο, πώς θα έχει συνταχθεί και ίσως η γραμματεία να μην, να μας στέλνει όλα τα κείμενα, να μας στέλνει μια σύνθεση, να μας στέλνει τα, τα προβληματικά σημεία, τα κυριότερα σημεία. Και εμείς ελπίζουμε να μπορέσουμε να επιφέρουμε διορθώσεις πριν από την έγκρισή τους, γιατί όταν, φτάνουμε, όταν φτάσουμε το Μάρτιο το παιχνίδι θα έχει τελειώσει. Εκεί ψηφίζουμε ναι ή όχι. Το κατάλαβαν όλοι. Και πάλι ο George. Ε, Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, όλη η δουλειά θα γίνει πριν το Μάρτιο, ώστε να δούμε ότι λαμβάνονται υπόψη, ε, να ληφθούν υπόψη τα, οι ανησυχίες μας. Αλλά και πάλι ανέκυπτο θέμα το κατά πόσο δικαιούνται λόγο ε, στους εμπειρογνώμονές μας δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα έχουν την πολιτική εντολή να επισημάνουν κάποιε διορθώσει που μπορεί να γίνουν στο κείμενο, λαμβάνοντα υπόψη τι ανησυχίε μα. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον Αγνιού, αλλά με συγχωρεί να πω κάτι στον Τζόρτζ. Πρέπει να ε, να μπορέσει το μέλος να εκφραστεί όσο το δυνατόν νωρίτερα σε περίπτωση που υπάρχει μια διαφορά. Ας μιλούμε για τα εγωπρόβατα. Το κάναμε και στην Ολομέλεια. Υπάρχει μια πολιτική συμφωνία, ε, θα πρέπει να, δο, να, δίδονται βοήθεια, να δίνεται βοήθεια για όλα τα ε, ζωικά είδη. ο εμπειρογνώμονάς μας εκεί μπορεί να μιλήσει, να πει επ' αυτού. Δεν έχει όμως πολιτική εντολή, δεν μπορεί να πει όχι κάνετε λάθος θα πρέπει βέβαια αμέσως να, αναφέρει τα θέματα στην Επιτροπή μας μέσω της συνάντησης των συντονιστών ή μέσω της συνεδρίασης της Επιτροπής μας και φυσικά εμείς θα κάνουμε τις παρατηρήσεις μας και θα τις στείλουμε ως πολιτικό μήνυμα ότι είμαστε κατά αυτής της ερμηνείας για παράδειγμα. Ε, πρόκειται για μια διαπραγμάτευση ε, μεταξύ των εθνικών εμπειρογνωμόνων και ημών. Ε, βέβαια, μπορεί να θίξει κάποια θέματα ερμηνείας, αλλά δεν μπορεί να μπει στην ουσία Γι' αυτό ακριβώς εμείς πρέπει να έχουμε μια στρατηγική, να μας ενημερώνουν οι εμπειρογνώμονες άμεσα και μετά στην συνέχεια να πούμε τις απόψεις μας και να πούμε στην Επιτροπή αν δεν το διορθώσετε θα το καταψηφίσουμε, θα το απορρίψουμε. Αγνιό. Νομίζω ότι η συζήτηση που μόλις είχαμε είναι απαραίτητε γνώσει για κάποιον που θέλει να γνωρίζει πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε σήμερα εσάς, τον Τζορτ Λάιν, τον κύριο από την Κομισιόν, που δεν μπορείτε να συμφωνήσετε για το ποιος έχει ποια εξουσία, πού και πότε. Ε, σίγουρα η ε, Επιτροπή Γεωργίας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να αναθέσει στον γραμματέα της να μιλήσει σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής και το γεγονός ότι αυτό συζητιέται αυτή τη στιγμή είναι πολύ περίεργο. Ευχαριστώ. <laughs> My friend. Uh, Φίλε μου, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, όπως είπε και ο Άγνιου. Ε, είναι σημαντικό και είναι αλήθεια ότι συζητούμε και στο πλαίσιο μιας άλλης επιτροπής πώς θα διαχειριστούμε τις κατεξουσιοδότης πράξη. Πρόκειται για την έκθεση Ζάιερ. Νομίζω ότι κάποιος θα το ξέρει. Στην έκθεση εκείνη το αντικείμενο είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να παρέμβει καλύτερα το Κοινοβούλιο στην εφαρμογή των κανονισμών μέσω των κατεξουσιοδότησης πράξεων. Θα γίνουν και προτάσεις. Υπάρχει και η πρόταση να ορίζεται εισηγητής. Κατανοείτε ότι είναι πολύ περίπλικα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να επιφορτήσουμε όλους τους συναδέλφους να παρακολουθούν τις κατεξουσιοδότησης πράξεις. Ε, ε, υπάρχει πρόβλεψη για 2.000 κατεξουσιοδότησης πράξεις ε, επί των τεσσάρων νομοθετικών ντοσιέ δεν ξέρω πόσες θα βγουν 12-14 κατεξουσιοδότης πράξης. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με κάθε κατεξουσιοδότης πράξη σαν να επρόκειτο για κάποια νομοθετική πράξη. Εφαρμοστική πράξη υποτίθεται ότι είναι. Θα πρέπει λοιπόν να χτίσουμε έναν μηχανισμό ελέγχου, παρακολούθησης και αν βλέπουμε κάτι ανησυχητικό αμέσως να λαμβάνουμε μια πολιτική απόφαση. Πρώτα μεταξύ των συντονιστών και μετά από την Επιτροπή. Ε, είναι, πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο ε, ακριβώς αυτή τη στιγμή συζητούμε. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω. Για άλλη μια στιγμή ότι η κατεξουσιοδότηση πράξη ε, δεν είναι και κάτι τραγικό αν δεν συμφωνήσουμε μαζί της, γιατί εν τέλει μπορούμε να την απορρίψουμε. Είμαστε, δικαιούμαστε να νομιμοποιούμαστε να απορρίψουμε. Λοιπόν, δεν θέλω να, να μην μεγενθύνουμε το, το ζήτημα. Είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστούμε, αλλά να μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Ε, θα πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό, να επηρεάζουμε, να διορθώνουμε τα σχέδια αυτά, αλλά εν τέλει αν το Κοινοβούλιο δεν είναι ικανοποιημένο από τις κατεξουσιδότητες πράξεις μπορεί ε, να την απορρίψει το Μάρτιο. Όταν λοιπόν ε, έρχονται μπροστά μας στην τελική τους μορφή τα κείμενα, τα κείμενα ε, μας ικανοποιούν, δεν μας ικανοποιούν. Μετά το Μάρτιο είτε δεχόμαστε είτε απορρίπτουμε. Τζιμ, θέλεις το λόγο, παρακαλώ. think we have Νομίζω ότι όταν η Κομισιόν ε, μιλά για εμπειρογνώμονα και είδαμε την Επιτροπή που ερχόταν ε, στους τριμερείς ε, διαλόγους και για κάθε παράγραφο που μιλάμε έχουν εμπειρογνώμονες. Εμείς εδώ στην Επιτροπή μας έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους αλλά δεν είναι εμπειρογνώμονες σε κάποιους τομείς. Η Επιτροπή ε, συγκεντρώνει ανθρώπους από τα διάφορα κρατημέλη και είναι πυρογνώμονες. Εμείς λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε ε, το, το τάδε ή το δίνα, αλλά ε, υπάρχουν τρόποι που δεν μπορεί να γίνει κάτι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με τι τρόπο θα εξετάζεται η δική μας συνεισφορά. Δεν λέω ότι είναι λάθος αυτά που κάνει η Επιτροπή, διότι Μπορεί να είναι λογικά κάποια από τα πράγματα που προτείνει, αλλά δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν με τέτοιο τρόπο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα βαθμό ευελιξίας για να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να αναγνωρίσουμε πού βρίσκεται το πρόβλημα. Θα πρέπει να εργαστούμε επικοδομητικά, αλλά και η Κομισιόν θα πρέπει να καταλάβει ότι έχουμε να παίξουμε κάποιο ρόλο και πώς θα παίξουμε τον ρόλο αυτόν. Και επίσης φαντάζομαι ότι τίθεται και ένα θέμα εμπιστευτικότητας εδώ. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Τζίμα. Θα έλεγα ότι αρκετά ε, ανατάμαμε το θέμα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έναν κατάλογο ε, σημείων. Θα μας βοηθήσει και το έγγραφο της GSA των 20 ε, Υπουργών στις 2 Δεκεμβρίου και κλεισμένων των θυρών θα συζητήσουμε με τους εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και το επιτελείο του Επιτρόπου για να δούμε τα υπέρ και τα κατά. Ευχαριστώ. Περνούμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης, επιλογή, φυτική επιλογή, επιλογές για την βελτίωση της ποιότητας και των αποδόσεων. Θα μιλήσουμε και για τα φυτικά γενετικά στοιχεία σε μια δημόσια ακρόαση. Αποφασίσαμε να καταρτήσουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Ε, ο κύριος Πόλσεν θα παρουσιάσει την έκθεσή του ε, για το θέμα αυτό. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας ε, συνεκτιμά τις μελλοντικές προκλήσεις του γεωργικού τομέα, την, ε, την γενετική βελτίωση των φυτών, και την, ε, το πώς θα θρέψουμε έναν αυξανόμενο πληθυσμό με, τον πεπερασμένο, με τους πεπερασμένους φυσικούς πόρους που διαθέτουμε. Υπάρχει εστίαση ε, στην τεχνολογία, ε, στη γενετική έρευνα και στους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις. Δίνω το λόγο στον κύριο Πόλσεν, στην κυρία Πόλσεν, με συγχωρείτε, και στη συνέχεια θα συζητήσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περιμένω να φορέσετε τα ακουστικά. Θα είμαι πάρα πάρα πολύ σύντομη όσον αφορά την αφετηρία της ε, του ε, σχεδίου έκθεσης πρωτοβουλίας μας. Το θέμα είναι ότι κατά 70% θα πρέπει να αυξηθεί ε, η συγκομιδή τροφίμων ε, τα επόμενα 30-40 έτη. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να αυξήσουμε το δυναμικό, δεν υπάρχει περισσότερη αρρώσιμη γη, του αντίον λιγότερη υπάρχει. Το νερό θα μοιράζεται με πιο άνισο τρόπο από ότι σήμερα. Μεγάλες ε, λοιπόν ε, αλλαγές μας περιμένουν ε, και τεράστιες προκλήσεις. Έχουμε επίσης το φαινόμενο ότι παγκοσμίω μειώνεται η συγκομιδή, όχι πάρα πολύ, έχει επιβρανθεί η πτώση, αλλά δεν αυξάνεται με τον τρόπο που αυξανόταν σε προηγούμενους αιώνες κάπως ε, καταστροφικό ε, όταν διαβάζει κανείς ε, τα σχετικά έγγραφα είναι ότι η ποικιλομορφία, η βιοπικιλότητα στην Γεωργία έχει μειωθεί κατά 75%. το, την τελευταία πεντηκονταετία και αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ. Ε, το συζητάμε αυτό συνέχεια, το συζητήσαμε και χθε ε, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την υγεία των ζώων. Υπάρχουν τόσο, μεγάλες, τόσο αλλαγές ε, ανάμεσα στην Βόρεια και την Νότια Ευρώπη, την Παράκτια και την Υπηρωτική. Ε, υπάρχει λοιπόν Χρειαζόμαστε μεγάλη βιοπικιλότητα στην Ευρώπη και για να αυξήσουμε τη συγκομιδή μας και για να διατηρήσουμε τις, τους παραδοσιακούς τρόπους ε, ζωής και γεωργίας. Ο τομέας βελτίωσης ε, των ε, φυτών περιορίζεται, συγκεντρώνεται σε έξι μεγάλες πολυεθνικές ε, εταιρείες οι οποίες ε, έχουν ε, δυσανάλογη εξουσία στον τομέα της γεωργίας. Εγώ θα ήθελα η Ευρώπη να τους πάρει αυτή την εξουσία, να την πάρει πίσω. Διότι αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποίησαν ε, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ε, για να πετύχουν ε, καλύτερη θρεπτική αξία και για τη διατήρηση της ποικιλομορφίας. Έχουν συγκεντρωθεί στην προσαρμογή των φυτών στα δικά τους ε, χημικά, κάτι που ε, αυξάνει το κέρδος της και βέβαια δεν είναι κακό μια εταιρεία να ε, αγωνίζεται για το κέρδος της, αλλά αυτό δεν συμπίπτει πάντα με τις ανάγκες της ανθρωπότητας και του κλίματος και, και του περιβάλλοντος. με τις ε, τεχνικές εξελίξεις ε, που είδαμε τα τελευταία 10-15 χρόνια, σήμερα ε, έχουμε μια σειρά διαφορετικών τεχνικών στη διάθεσή μας που μοιάζουν με τις τεχνικές γενετικής τροποποίησης που δεν καλύπτονται όμως από την παρούσα νομοθεσία και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους Όταν σπέρνουμε λοιπόν ναι, καρότα ή ε, κουνουπίδια σήμερα, δεν ε, μπορούμε ε, να διαπιστώσουμε από, με τι τεχνικές έχουν παραχθεί οι σπόροι αυτοί. Προσπαθώ λοιπόν να πω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία, νέα και παλαιά, σε όλο τον κόσμο αλλά και στις τοπικές κοινότητες στην Ευρώπη, και γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να διεξάγει έρευνα και να έχουμε ε, έναν πλήρη και εντελεχή διάλογο σχετικά με το πού βρισκόμαστε σήμερα, ποιες θα είναι οι ανάγκες μας ε, στο μέλλον, πώς θα χειριστούμε την ε, πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Ουσιαστικά απλά προσπάθησα να θέσω μια σειρά εφιών ερωτήσεων δεν μπορώ όμως να ισχυριστώ ότι έχω απαντήσεις στο σχέδιο έκθεσής μου στην έκθεση πρωτοβουλίας. Για να έχουμε όμως τις σωστές απαντήσεις, πιστεύω ότι θα πρέπει να διατυπώσουμε σωστά και με εγνωσμένο τρόπο τις ερωτήσεις μας στην Επιτροπή Γεωργίας, ε, λοιπόν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς, εμείς ειλικρινά εμείς έχουμε την πολιτική και ε, ηθική ευθύνη για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις για να χειριστούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η πολιτική γεωργίας είναι ευρωπαϊκή πολιτική και σε περιορισμένο βαθμό είναι εθνική πολιτική.

σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, σε έναν κόσμο όπου οι πόροι συνεχώς μειώνονται. Ε, βασίζομαι στην βοήθειά σας ε, για να μπορέσουμε μαζί να διατυπώσουμε σωστές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Μάριτ. Ξεκινούμε την συζήτηση. Τέσσερις συνάδελφοι. Ο κύριος Καλινόσκη πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μάρτ Πάρσεν γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεσή της και είναι ενδιαφέρουσα γιατί το θέμα αυτό είναι συναρπαστικό πραγματικά. Πώς θα εξασφαλίσουμε ε, τρόφιμα για την ανθρωπότητα όταν οι ανάγκες τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν κατά 70% και ίσως και περισσότερο. Ενώ έχουμε συγκεκριμένους περιορισμούς και αυτούς ανέλησε και μας περιέγραψε η εισηγήτρια περιορισμός των αρρώσιμων καλλιεργειών, αλλά και πεπερασμένου υδάτινου σπόρους. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν θεμελιώδη σημασία. Πώ θα ανταποκριθούμε λοιπόν σε αυτές τι τεράστιε προκλήσεις δεδομένων αυτών των περιορισμών που αντιμετωπίζουμε, χάρη στην επιστήμη, χάρη στην έρευνα. Χρειαζόμαστε λοιπόν την επιστήμη και την έρευνα, αλλά έχουμε και παράλληλους στόχους στη διασφάλιση της ε, βιοπικιλότητας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και αυτά θα πρέπει να τα Έχω λοιπόν μια ερώτηση προς ε, την κυρία εισηγητρία γιατί μάλλον δεν κατάλαβα καλά ένα σημείο. Για το σημείο 6 συγκεκριμένα της ε, έκθεσής σας που λέτε ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε, στις διάφορες τεχνολογίες στις προσιτές τεχνολογίες. Τι εννοείται προσιτές τεχνολογίες, δηλαδή πρόσβαση και στις τεχνολογίες ε, ε γενετικής ε, τροποποίησης, ε, γιατί κατά τη γνώμη μου θα πρέπει αυτές τις νέες τεχνολογίες στην Ευρώπη να συνυπάρχουν με τις υπάρχουσες, αλλά με στόχο να διασφαλίσουμε την βιοπικιλότητα. Επίσης εκφράζετε τη θλίψη σας για την αδεσπόσα θέση μερικών μεγάλων πολυεθνικών. Έχετε δίκιο, αυτό ισχύει. Απ' την άλλη όμως λέτε ότι είναι πολύ δαπανηρή καλλιέργεια νέων ποικιλιών. Ιδιαίτερα όταν δεν έχουμε μηχανισμούς που στηρίζουν την έρευνα. Γι' αυτό και η θέση, η κατάσταση αυτή ευνοεί περισσότερο τις μεγάλες πολυεθνικές ε, Γι' αυτό θα ήθελα να, απευθύνω έκκληση ώστε να εξασφαλίσουμε κατάλληλη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προβλέψουμε μηχανισμούς που θα μπορέσουν μακροπρόθεσμα να στηρίξουν την, επιστημονική, την ευρωπαϊκή επιστήμη και την ευρωπαϊκή έρευνα. Γιατί ε, ή αλλιώς θα παραμείνει ε, ευσεβής πόθος αυτή η επιθυμία για ε, να περιορίσουμε τη δεσπόσα θέση μερικών μεγάλων πολυεθνικών. Αν δεν προβλέψουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση, ό,τι και να λέμε θα συνεχίσουν αυτές οι μεγάλες ε, πολυεθνικές να καρπώνουν ουσιαστικά όλη την αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καλινόφσκι. Λεμπρόν και στη συνέχεια Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μάριτ Πόλσεν για την ε, πολύ καλή εργασία της ε, και την ανάλυση κατάστασης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ε, γεωργίας. Είναι αρκετά εξαντλητική η ανάλυση που κάνει, δελεχέστατη και ευτυχώς αποφεύγει και το δογματισμό των περιρέοντα που πολύ συχνά στις περιπτώσεις αυτές εμποδίζει την σωστή διάγνωση και ανάλυση θολώνει και τη σκέψη αλλά και την ποιότητα των προτάσεων. Πολύ ε, ενδιαφέρουσα στην έκθεσή της είναι η άποψη ότι είναι εξίσου σημαντική η επισήμαση της ανάγκης ε, παραγωγής νέων ειδών και ποικιλιών για να ανταποκριθούμε στην ε, δραστική αύξηση των παγκόσμιων αναγκών των επιστημιστικών, ενώ ταυτόχρονα έχουμε κλιματικές αλλαγές, έχουμε ε, αλλαγές που προκύπτουν από διάφορες ε, ασθένειες, κάτι που τροποποιεί το γενικό κλίμα και επίσης επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας νέων ειδών, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνεται και διατρανώνεται την ανάγκη της διασφάλισης του γενετικού υλικού, της γενετικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα διαφύλαξη των τοπικών και περιφερειακών ποικιλιών και ειδών. Εγώ δίνω μάχη για να προασπίσουμε μια ε, τοπική ποικιλία φρέσκου κρεμμυδιού και πραγματικά είναι δύσκολο από τη μια να ενισχύσουμε την ανάπτυξη ε, και ταυτόχρονα να προωθήσουμε και να προαγάγουμε και τα παραδοσιακά μας ε, ήδη. Ενώ εσείς ε, φαίνεται ότι ήρθατε μια ισορροπημένη πρόταση. Επίσης, ε, για την ανάπτυξη, ο δρόμος που χρησιμοποιείται είναι σωστός γιατί πολλές φορές υπάρχει μεγάλος διαχωρισμός. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια ε, φιλόδοξη στρατηγική για τα φυτικά είδη, συνεκτική, που θα αποδέχεται την ανάγκη της διαφοροποίησης των διαφόρων παραγόντων ναι, ναι, βέβαια, θα έχουμε και τις μεγάλες εταιρείες. Εγώ δεν καταγγέλω τη μονοπωλιακή ε, στρατηγική, γιατί δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Αυτό καταγγέλλεται μια τέτοια μονοπωλιακή στρατηγική. Ε, γι' αυτό και χρειαζόμαστε ελέγχους. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε και τα τοπικά ερευνητικά κέντρα, γιατί πραγματικά είναι πολύ, έχουν σημαντικό δυναμικό. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε τους πόρους ώστε να μπορέσουν αυτά τα τοπικά ερευνητικά κέντρα να εκτελέσουν ε, τις εργασίες τους και μάλιστα θα πρέπει να έχουν και ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τουλάχιστον μία δεκαετία για να είναι ασφαλής. Έλεγχος λοιπόν, χρηματοοικονομική ενίσχυση και μία βιωσιμότητα. Πολύ καλές οι βάσεις της πρότασης αυτής, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα να κάνουμε περισσότερο ένα απολογισμό της κατάστασης, όχι μόνο ένα ευχολόγιο. Ε, είναι πολύ ε, αξιέπαινη έκθεση γιατί πραγματικά ανοίγει τις πόρτες σε πολλές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ανιές. Λουίς Κάπολα Σάντος. Στη συνέχεια Άγνιο. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να σε την κυρία Πόλσεν ε, για το έργο της. Γιατί πραγματικά ταράζει τα νερά σε ένα πρόβλημα που είναι πραγματικά αδύνατο να το, να για το οποίο είναι αδύνατο να διαφορήσει κανείς. Είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να διαφεύγει της προσοχής μας. Ένα από τα αδιαφυσβήτητα θέματα στα, όταν συζητούμε για κάτι τέτοιο, το θέμα της βιοτεχνολογίας που πολύ επιδέξει αποφεύγει η κυρία Πόλσεν. Πιστεύω ότι σε αυτή τη συζήτηση δεν θα πρέπει να έχουμε ούτε προκαταλήψεις ούτε ταμπού και να αναλύουμε όλε τι πτυχέ αυτού του θέματος, συμπεριλαμβάνοντα και την βιοτεχνολογία. Επίση, με όλα τα στοιχεία που μα δίνει πραγματικά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου γιατί αναφέρει ότι τον 20ο αιώνα χάσαμε το 75% τη ε, φυτική βιοπικιλότητα. Είναι τραγικό, δημιουργεί τεράστιες ανησυχίες και πριν από μερικούς μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθήσαμε μία παρουσίαση που μας είπε ότι η ε, αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα χρειάζεται μία ε, ε, έκταση αντίστοιχη με της Αφρικής για να παράγει φυτικά είδη και αντίστοιχη για της Νοτιού Αμερικής για, να, για την κτηνοτροφία. Δεδομένου όμως και των δημογραφικών περιορισμών θα πρέπει στον 21ο αιώνα να βρούμε λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Μία από τις λύσεις είναι η βελτίωση των ποικιλιών φυσικά του φυτικού κόσμου, αλλά και η διερεύνηση άλλων λύσεων που θα προκύψουν από την επιστήμη και από την έρευνα. Και αυτό το θέμα πολύ σωστά αναφέρεται στην έκθεση της κυρίας Πόλσεν και πολύ εύστοχα. Τη συγχαίρω λοιπόν για το έργο της Είμαι σίγουρος ότι είναι σημαντικός συναγερμός ε, αυτή η έκθεση και αυτή την προειδοποίηση θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αναζητήσουμε λύσεις για ένα πρόβλημα που τις επόμενες δεκαετίες θα γίνει το μείζον πρόβλημα της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ. Όντως. Άγνιο και μετά ο Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την, την κυρία Πόλσον που τουλάχιστον επισήμανε αυτά τα θέματα. Ακόμη και αν δεν συμφωνώ μαζί τη ε, για τα σημεία αυτά. Εγώ θα μιλήσω για την ταπεινή πατάτα. Ε, ένα τρόφιμο που το καταναλώνουμε παντού σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι δυσδυτικό είδο, γιατί ανακαλύφθηκε στην Αμερική, μεταφέρθηκε εδώ και μετά ξανα ε, βρέθηκε πριν από 170 ε, χρόνια, αλλά είχαμε ένα, μια μεγάλη επιδημία, ε, οπότε είχαμε και μιλιμοκτονία στην ε, Ιρλανδία. Τότε οι πυρογνώμονες μας, οι τεχνικοί, ανέπτυξαν για το παράσιτο αυτό παρασιτοκτόνα για να το εξολοθρεύσουν, αλλά δυστυχώς είναι μια παθογόνος ουσία αυτό το παράσιτο ε, πολύ ε, επίμονο και επανερχόταν παρά τα παρασιτοκτόνα που επινόησαν οι επιστήμονες την τελευταία, ε, τον τελευταίο αιώνα. Και μάλιστα δεν απειλείται μόνο τα φύλλα αλλά και το βολβό αυτό το ζυζάνιο. είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Τώρα φτάσαμε σε μια κατάσταση που μπορεί κανείς μόνο 19 εντό εισαγωγικών ε, φορές να ψεκάσει μέσα σε μία εποχή, αλλά όσο περνά τα χρόνια, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείε που δεν είναι τις αρισκές κυρίες Πάουσεν συστηματικά παρήγαν όλο και πιο ε, ακριβές λύσεις, γιατί η χημία, οι χημική διαδικασία είναι πολύ πιο περίπλοκες, αλλά φαίνεται ότι εξακολουθούμε να χάνουμε την ε, μάχη. 30 μίλια από το δικό μου σπίτι υπάρχει ένα ερευνητικό κέντρο και στο ερευνητικό αυτό κέντρο βρέθηκε η λύση. Πήγα να τη δω. Και το πρώτο πράγμα που με κατέπληξε είναι ότι χρειάστηκε να ξοδέψουν 20.000 ε, λίρες για να ε, σηκώσουν ε, φραγμούς για να κάνουν φράχτες για να αποτρέψουν τους ακτιβιστές να έρθουν και να καταστρέψουν αυτά που είχαν εφεύρει. Χρησιμοποίησαν τη βιοτεχνολογία για τη γενετική μηχανική να βρουν ένα γονίδιο από ένα φυτό που ήδη υπάρχει στην Νότια Αμερική που είναι, είναι σαν την πατάτα και είναι ανθεκτικό σε αυτό το παράσιτο, σε αυτό το ζυζάνιο. Και κατάφεραν από αυτό το μη βρόσιμο φυτό να πάνε αυτό το γονίδιο και να το εισαγάγουν στην ε, βασική ποικιλία της πατάτας. Θα θεωρούσε κανείς ότι θα ήταν... Ε, ε, θα, θα είχαν αυτή η λύση. Αλλά τελικά διαπίστωσαν οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν είχαν αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναφαδόν κατά της ε, γενετικής ε, τροποποίησης. Ε, δεν την επιτρέπει παρά το γεγονός ότι αυτή η μέθοδος η μετάλλαξη δίνει λύσεις και έτσι αποθαρρύνουμε επιστήμονες που έχουν λύσεις από το να κάνουν τις έρευνες. Πώς λοιπόν θα αντιδράσουν αυτοί οι επιστήμονες, είτε θα φύγουν στην Αλοδαπή, όπου το έργο τους ε, αξιολογείται καλύτερα, εκτιμάται καλύτερα και προωθείται ή θα πούν «Α, οι πράσινοι ε, ακτιβιστές ε, δεν επιδοκίμασαν την τελευταία μας λύση, γιατί λοιπόν να πουμε στον κόπο να επινοήσουμε νέα». Ευχαριστώ κύριος Ντόρφμαν και μετά κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αδιαμφισβήτητα η αντιμετώπιση του θέματος πώς στο μέλλον θα ταΐσουμε τον κόσμο ε, στο μέλλον. Ε, στο ερώτημα αυτό παίζει διαφυσβήτηκα μεγάλο ρόλο ε, η φυτική παραγωγή. Και στο παρελθόν κοιτάζαμε επικριτικά τις γεωργικές πρακτικές. Για παράδειγμα πριν 100 χρόνια υπήρχε περονόσπορος ε, στην Ευρώπη και θεωρήθηκε τότε ότι αυτό σχετιζόταν με, την, με τις νέες πρακτικές στον τομέα του ίνου. Πάντα λοιπόν ε, εξεταζόταν πάντα επικριτικά η φυτική παραγωγή. Κυρία Πάουλσεν. Γράφεται εδώ ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με την φυτική παραγωγή. Σπάνια συμφωνώ με τον ε, συνάδελφο Άγνιου, αλλά θα συμφωνήσω τώρα. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν για αυτό. Είναι αυτονόητο ότι μια εταιρεία που ασχολείται με την φυτική παραγωγή ότι τουλάχιστον οι μεγάλες ε, ε, εταιρείες ε, θέλουν τα προϊόντα που αναπτύσσουν να μπορούν να τα απολούν οι ίδιοι σε όλο τον κόσμο. Στο σημείο 14 της έκθεσης ξεκινάει ο λαϊκισμός. Οι μεγάλη είναι η κακή και οι μικρή είναι οι καλή. Πού το γράφει αυτό. Μήπως ε, πρέπει να, ε, ε, να εκπονηθεί ένα έγγραφο όπου να φαίνεται ποια είναι η δομή της φυτικής παραγωγής στην Ευρώπη. Υπάρχουν χιλιάδες παραγωγή χιλιάδες μικροί παραγωγή που ασχολούνται με λιγότερο σημαντικές καλλιέργειες εντό εισαγωγικών, τα διαφόρων ειδών λαχανικά κλπ. Ε, στην Ευρώπη λοιπόν αυτοί κινούνται σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο. Και στο 20 δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε τόσο απλά να λέμε ότι δεν εμφανίζονται νέα είδη. Κοιτάξτε μια εφημερίδα που να απευθύνεται σε σε πόσα νέα είδη παράγονται κάθε χρόνο. Λυπάμαι κυρία Πόλσεν, αλλά πρέπει να επικρίνω την έκθεση αυτή. Αν ε, θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι ο τομέα σήμερα στην Ευρώπη, ποιο εργάζεται εδώ, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη και όχι απλά να λέμε ότι οι μεγάλοι είναι κακοί και καταστρέφουν τη βιοπικιλότητα ενώ οι μικροί είναι καλοί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι εταιρείες εργάζονται στην Ευρώπη, πώς μπορούμε να συμβάλλουμε ε, ε, στη βελτίωση της κατάστασης στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να μην συμφωνεί κανείς με την εισηγήτρια. Μαρτίν Πόλσεν Κύριε Πόλσεν, σας ευχαριστούμε για την έκθεση αυτή. Υπάρχουν πολλά θέματα εδώ που θέλω ε, να στηρίξω. Δεν έχω καμία ε, αντίρρηση στην έρευνα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ότι η έρευνα αυτή κατευθύνεται από τους μεγάλους εντό εισαγωγικών ε, και κατευθύνεται σε προσκεκριμένη κατεύθυνση. κατεύθυνση. Τα τελευταία χρόνια Ε, είδαμε ότι χρηματοδοτούνται οι έρευνες από, αυτού από αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν μετά τα αποτελέσματα της έρευνας, ε, αλλά ε, αυτό εντάξει, αλλά αυτό γίνεται σε τομείς που μπορεί να βγάλει κανείς πολλά χρήματα. Για παράδειγμα, Βλέπουμε ότι ε, χρηματοδοτούνται πολλές ε, έρευνες ε, για το καλαπόκι και το στάρι, αλλά όχι για άλλα φυτά τα οποία δεν είναι τόσο επικερδή. Είπατε ότι πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή κατά 70%. Δεν... Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην έρευνα. Ε, με αυτά που παράγουμε ε, στον κόσμο μπορούμε να ταΐσουμε 12, εκατομμύρια, 12 δισεκατομμύρια ανθρώπους, αλλά είναι θέμα ε, κατανομής και το 50% των τροφίμων στην Ευρώπη, στον πολιτισμένο κόσμο, στον αναπτυγμένο κόσμο, τα πετάμε στα σκουπίδια οι υποδομές ε, μεταφορών ε, δεν, δεν αρκούν ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα τρόφιμα αυτά προς τους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Να λέμε ότι ναι, πρέπει να ξανασκεφτούμε ε, την γενετική τροποποίηση. Ε, ζήτω συγγνώμη, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Και αναφέρθηκαν οι πατάτες, αλλά αυτό είναι πρόβλημα των μονοκαλλιεργιών ε, και τέτοια προβλήματα ε, ε, υπάρχουν παντού και παντού διαπιστώνονται. Λέμε λοιπόν, ωραία, αν προσθέσουμε και λίγη γενετική τεχνική θα βελτιωθεί η κατάσταση της μονοκαλλιέργειας. Όχι. Θέλουμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα του εδάφους, ε, παρότι ο κύριος ε, Άγνιου μπορεί να διαφωνεί, αλλά έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν. Ε, δεν αρκεί λοιπόν απλά η γενετική τεχνική για να βελτιωθεί η κατάσταση. Το απόγευμα έχουμε την έκθεση Σιλβέστρης για τα, τους σπόρους. εγώ ανησυχώ ότι με την προσέγγιση αυτή δεν αντιμετωπίζουμε ακριβώς ε, τα προβλήματα που έχουμε στον τομέα της βιοπικιλότητα, αλλά ακολουθούμε την κατεύθυνση που έχουν ακολουθήσει οι μεγάλες εταιρείε μέχρι τώρα, ότι επικεντρωνόμαστε σε κάποια, σε σημαντικά μερίδια στην αγορά. Θα πρέπει λοιπόν ε, η πολιτική, εμείς να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ε, χρειαζόμαστε ε, είδη, φυτικά είδη τα οποία ε, είναι προσαρμοσμένα στην αλλαγή του κλίματος. αλλά θα πρέπει να δούμε προς ποια κατεύθυνση κινείται ο κύριος Σιλβέστης με την εκθεσή του. Προωθούμε τα μονοπόλια. ή πράγματι ε, προωθούμε τη βιοπικιλότητα. Εγώ ανησυχώ. ότι η έκθεση Σιλβέστρης δεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Κυρία Μακιντάιρ και μετά ζήτησε το λόγο για λίγο ο κύριος Αλμπερντές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Πόλσεν ε, θερμά για την έκθεσή της, γιατί το θέμα πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό να αυξήσουμε και την ποιότητα, αλλά πρώτα απ' όλα την, ε, τις οδηγές, την αποδοτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται 10 χρόνια για την ανάπτυξη μιας νέας ποικιλία σπόρων μας, λέει η κυρία Πόλσεν. Σε ό,τι αφορά την, αύξηση την ανάπτυξη χορτονομής, χρειάζεται 18 χρόνια. Ε, οπότε θα πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τις τεχνικές μας ε, ε, και φυσικά υπάρχουν μερικές τεχνικές που επιταχύνουν την βλάστηση, και είναι κρίμα, ή μάλλον την ε, καλλιέργεια των νέων ποικιλιών. Και κρίμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάθετα οποιασδήποτε, κατά οποιασδήποτε μορφής γενετικής μηχανικής. Γιατί πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε πλήρως το θέμα. Ε, να έχουμε μια εμπεριστατωμένη γνώμη και όχι απλώς ε, να απορρίπτουμε όλο όλος χερός οποιαδήποτε προσέγγιση της γενετικής μετάλλαξης. Τα θέματα των απορκευτικών είναι πολύ σημαντικά. Όταν μιλούμε για αύξηση τη ε, σοδιά ε, συγκεκριμένων ε, αρρώσιμων καλλιεργιών, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το 18% τη συνολική αξία τη γεωργική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται μόνο από 3% των αρρώσιμων καλλιεργιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αρρώσιμων γεών. Οπότε υπάρχει δυνατότητα να αυξήσουμε την απόδοση των καλλιεργιών απορροκυπευτικών και να έχουμε και τεράστια ωφέλη για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη αντικατάσταση των εισαγωγών μας αν επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στα απορροκυπευτικά μας. Διαφωνώ με μερικά σημεία της έκθεσης. Μερικά τα ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κυρίως το θέμα της χρήσης των μυκητοκτόνων, φυτοκτόνων, παρασιτοκτόνων και κάποιων χημικών ουσιών που αρχίζουμε να παγορεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συνεχίζουμε παρόλα αυτά να εισαγάγουμε απορροκυπευτικά από άλλες περιοχές του κόσμου όπου επιτρέπονται τέτοιου είδους ε, φυτοφάρμακα. Οπότε δένουμε τα χέρια πισόπλατα πίσω από την πλάτη των ε, γεωργών μας. Τους φέρνουμε σε πολύ δύσκολη θέση και σε μειονεκτική θέση, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε τις εισαγωγές από χώρε που εφαρμόζουν και χρησιμοποιούν προϊόντα που εμείς απαγορεύουμε. Ενώ ταυτόχρονα μας ενδιαφέρει το θέμα της αύξησης αποδοτικότητας των εσοδιών μας δεν αρκεί απλώ να επιτίθεται τις μεγάλες εταιρείε. Είναι αναμφίβολο ότι και μικρές εταιρείε κάνουν, επιτελούν σημαντικό έργο, γιατί ιδιαίτερα στη δική μου πατρίδα και στη δική μου περιφέρεια έχουμε σημαντικό έργο των μικρών εταιριών. Θα ήθελα λοιπόν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Πάντως ευχαριστώ, ευχαριστώ την κυρία Πόλσεν, γιατί αν μη τι άλλο ε, έφερε στο επίκεντρο της συζήτησης αυτό το θέμα. Ευχαριστώ για την προεργασία της και θα καταθέσω και τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Μάκιν Τάιρε. Δες πρώτα και μετά Νταντέν. Ευχαριστώ Παύλο. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή που, η οποία σίγουρα θα μας οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ελπίζω στο τέλος να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή γραμμή. Ε, αλλά πήρα το λόγο λόγω του συναδέρφου Μάρτιν Χόισλινγκ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Μάρτιν το εξή σχετικά με τις ε, μονοκαλλιέργειες ε, στην ε, περιοχή μου. Παράγονται λίγες πατάτες μόνο για ιδία χρήση 0,1 εκτάρια, 0,2 εκτάρια, 0,3 εκτάρια. Αλλά όλοι αντιμετωπίζουμε το θέμα της συγκεκριμένης ασθένειας. Και Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η, ε, οι γεωργοί γιατί χρησιμοποιούν ε, χαλκό ε, η βιολογική η που είναι ε, πολύ δηλητηριώδης. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα και στην βιολογική παραγωγή. Δεν είναι μόνο η μονοκαλλιέργεια πρόβλημα. Η γεωργική ε, έρευνα στην Ευρώπη, αν δεν είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, θα οδηγήσει σε έξοδο των ερευνητών από την ε, Ευρώπη. Και και εγώ νιώθω καλά όταν αγοράζω από πολυεθνική ε, ε, ένα αυτοκίνητο, ένα Volkswagen ή κάτι τέτοιο. Ε, υπάρχουν ακόμα χειροποίητα αυτοκίνητα, αλλά μπορεί να μην έχω λεφτά για κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό αγοράζω από πολυεθνική εταιρεία αυτοκίνητο, διότι έχω τα λεφτά για κάτι τέτοιο. Grazie Alberto, Ευχαριστώ. Όταν μιλούμε για ε, βιοτέχνε ή μικρή ε, ε, εμβέλειας παραγωγού. φαντάζομαι δεν νοούσε την Πεζό ο κύριος Δες, που είναι σημαντικό παραγωγό και έχει και στην Αλσατή εργοστάσιο. Προσοχή στην επιλογή της, του κλάδου των φυτικών ειδών. Να έχουμε τις καλύτερες παραγωγικότητες και αυτό πετύχαμε τα τελευταία 70 χρόνια. Χάρη σε αυτούς τους τομείς λοιπόν ε, δεν μας απασχολεί πια το επιστηστικό θέμα τουλάχιστον ένα μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας παρόλο που για οικονομικούς λόγους το θέμα της επιστηστικής ασφάλειας ε, εξακολουθεί να προβληματίζει πολλούς. Τώρα, σε σχέση με τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, θέρμανσης του πλανήτη, για παράδειγμα, των ε, θερμικών ε, σοκ. Χρειαζόμαστε την έρευνα και κυρίως την έρευνα για τις ποικιλίε για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Και αν δεν στηρίξουμε αυτή την έρευνα θα είναι μεγάλο λάθος. Θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Βέβαια υπάρχει και ένα πολιτικό θέμα. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια και πώς θα αξιοποιήσουμε τα ερευνητικά απορίσματα. Εκεί έχουμε μια πολιτική επέμβαση που θα πρέπει να κάνουμε πρόσβαση σε όλους τους ερευνητές σε ό,τι φορά την ποικιλία του υπάρχοντος γενετικού υλικού. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή την πρόταση, πρόσβαση και να φροντίσουμε ώστε η βιοπικιλότητα που εξακολουθεί να αποτελεί καταπληκτικό γονιδιακό δυναμικό δεν θα πρέπει να είναι το προνόμιο ορισμένων μόνο. Δεν θα πρέπει να τις φετερίζονται λίγοι μόνο ερευνητές. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση όλων των ερευνητών στο γενετικό υλικό που υπάρχει στη διάθεσή μας. Τα σημεία 6 και 7, επίσης 14, 15 και 16 είναι κάπως περιοριστικά. Έχουμε στην Ευρώπη έναν τομέα έρευνας ε, για τις ποικιλίε των φυτών που δεν ανήκει στα χέρια των μεγάλων πολυεθνικών και αυτός ο τομέας ε, κάθε χρόνο ε, συμβάλλει στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Θα σας δώσω ένα μόνο αριθμητικό στοιχείο. Στη δική μου πατρίδα πέρυσι οι εξαγωγές διαφόρων ποικιλιών ε, σπόρων ε, αντιστοιχούσαν στο, σε 21 Airbus. Το να εξάγει κανείς 21 Airbus αεροπλάνα. Φυσικά δεν ε, εμφανίζει τους πηχαίους τίτλους ε, των εφημερίδων. Παρόλα αυτά είναι η πολύ σημαντική επίδοση του τομέα των ποικιλιών σε μία μόνο χώρα. Μιλάω μόνο για την Γαλλία. Οπότε έχουμε ένα σημαντικό τομέα που θα πρέπει να διαφυλάξουμε. Αν δεν αφήσουμε όμως την ευρωπαϊκή έρευνα να αναπτυχθεί όπως ε, θεωρούν απαραίτητοι επιστήμονες για να συνεχίσουμε ε, να έχουμε μια παρουσία στον κόσμο, θα βρεθούμε στο μέλλον να είμαστε εχμάλωτοι όμοιροι λίγων ε, αμερικανικών ομίλων. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τον τομέα της Ευρώπης για την παραγωγή ποικιλιών σπόρων. Ευχαριστώ Μισελ. Άγνιο και ο Μάρτιν θέλει να πάρει το λόγο και πάλι. Άγνιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο να, διευ... δευτερολογήσω μετά τις επιθώσεις που μου έκαναν κάποιοι για τον περονόσπορο της πατάτας. Ε, ε, είπα ότι συνδέεται με τη μονοκαλλιέργεια. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι μονοκαλλιέργεια οι πατάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι περισσότεροι που καλλιεργούν πατάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν 5-6 ε, χρόνια διαφορά και μάλιστα δεν το κάνουν εξαιτία του περονόσπορου της πατάτας, αλλά εξαιτία ε, μιας ασθένειας του εδάφους που κάθε πέντε χρόνια εξαφανίζεται. Γι' αυτό και προβλέπουν οι γεωργοί μας ε, διαστήματα πενταετή. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση μονοκαλλιέργεια τη πατάτας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ο περονόσπορος της πατάτας ε, οφείλεται σε καιρικέ συνθήκε. όταν ταυτόχρονα η υγρασία και η θερμοκρασία περνούν ένα συγκεκριμένο κατόφλι. Ε, σε 24-48 ώρες ε, όταν πληρούνται οι συνθήκες αυτές αυξάνεται, πολλαπλασιάζεται με εντυπωσιακό τρόπο ο περονόσπορος. Οπότε με την θέρμανση του πλανήτη ε, κανονικά θα σταματήσει ο περονόσπορος γιατί δεν θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για το πολλαπλασιασμό. Θα πρέπει λοιπόν να σταματούν οι πράσινοι ακτιβιστές να μας κατηγορούν για αυτά τα θέματα και να μας παραπλανούν με λαθασμένες πληροφορίες. Ο Άλμπερτ δυστυχώ ε, βγήκε από την αίθουσα, αλλά ε, δεν ανήκει στα βαρέα μέταλλα ο χαλκός. Ε, μήπως μπορείς να του το πεις ότι άλλα είναι τα βαρέα μέταλλα. Αλλά και σε άλλους τομείς χρησιμοποιείται ο χαλκός, για παράδειγμα, ε, στον ίνο χρησιμοποιούνται, στα μπέλια χρησιμοποιείται περισσότερο, περισσότερος χαλκός στις ε, μη οικολογικές από τις οικολογικές εκμεταλλεύσεις. Εγώ ίδιος ε, έχω καλλιεργήσει πατάτες, δεν είναι ότι δεν έχω καμία ιδέα για τον τομέα αυτό, αλλά ήταν πρόβλημα ότι ε, επιλέγει κανείς ε, μια καλλιέργεια και ε, αν επέλθει η καταστροφή δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. ο περιορισμός της ποικιλία. και είτε μιλάμε για ζώα είτε μιλάμε για φυτά, πολύ σύντομα γίνεται κανείς ευάλωτος και γι' αυτό και το κάνει αυτό κάθε οικολογική εκμετάλλευση. Φροντίζει να έχει ένα ευρύ φάσμα ειδών ώστε να μην εξαρτάται από μία ποικιλία. Υπάρχουν ε, κίνδυνοι εδώ και το θέμα είναι και οι πολυεθνικές ε, εταιρείε. Η Μονσάντο δεν είναι ε, γεωργική επιχείρηση, είναι χημικά. Και ε, ε γι' αυτό επενδύουν τόσα στι έρευνε, επειδή θέλουν να το συνδέσουν αυτό με τα χημικά τους. Θέλουν να πολλούν δηλαδή τους σπόρους μαζί με τα φυτοφάρμακα ως πακέτο. Αν κοιτάξει λοιπόν κανείς τις απώλειες ε, στην Ευρώπη που είχαμε θα διαπιστώσουμε ότι ε, χάνουμε ε, τις μικρές επιχειρήσεις ή αυτές εξαγοράζονται από τις μεγάλες και πρέπει να ακολουθήσουν τη στρατηγική τους. αυτό είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Επιτροπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε κάποιον από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας, Άιβι Corpy, ε, την κυρία Άιβερ Manor είναι εδώ. Έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Πόλσεν που έθιξε όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα για τις φυτικές ποικιλίε, την αναπαραγωγή των φυτών και την το θέμα της διατροφικής ασφάλειας ε, στον 21ο αιώνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια παγκόσμια ευθύνη πάνω σε αυτό, καθώς είναι παραγωγός σπόρων, ε, είναι ηγετική δύναμη στις εξαγωγές σπόρων και έχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στον τομέα. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή και όλοι συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σχετικά με την απώλεια της βιοπικιλότητας ε, ε, ε, μειώνεται η βιοπικιλότητα στα γεωργικά εδάφη γιατί χρησιμοποιούνται λιγότερα φυτικά είδη. Αν δείτε τα τρόφιμα που καταναλώνουμε θα δείτε ότι υπάρχουν περίπου 60 καλλιέργειες που στην Ευρώπη και αυτό που καταναλώνουμε είναι ένας περιορισμένος αριθμός καλλιεργιών, καλλιεργούμενων προϊόντων. Ε, λοιπόν, η μείωση αυτή ε, συμβαίνει στο επίπεδο των καλλιεργούμενων φυτών, η μείωση της βιοπικιλότητας. Ε, οι γενετικοί πόροι έχουν μεγάλη σημασία για την αναπαραγωγή των φυτών. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε, να διαφυλάξουμε τους γενετικούς πόρους ε, στη φύτευση, ναι, στα, δίκτυα και να υπάρχει πρόσβαση στους ε, γενετικούς πόρους σε ολόκληρον τον κόσμο. Γιατί από εκεί αντλούν ε, οι εταιρείε αναπαραγωγής φυτών το υλικό τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και υπάρχει μια διεθνή συνθήκη για τους γενετικούς πόρους και τη χρήση τους στη γεωργία. Για το θέμα της σπάνης, της σπάνης των πόρων, Υπάρχουν φόβοι ότι λόγω της ε, αλλαγής του κλίματος ε, θα υπάρχει λιγότερο διαθέσιμο νερό και άρα λιγότερες θρεπτικές ουσίες για τα φυτά, θα αναπτυχθούν νέες ασθένειες των φυτών και γι' αυτό είναι σημαντικό στις φυτικές μας ποικιλίε να χρησιμοποιούμε νέες να βρεθούν νέες βελτιωμένες ποικιλίε. Όταν αναπτύσσονται οι ποικιλίε αυτές θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε ανεξάρτητους ελέγχους και αξιόπιστους ελέγχους. Η Νομική Επιτροπή ε, έχει μια πρόταση ε, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να καθοδηγήσουμε την αναπαραγωγή των φυτών σε μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση, έτσι ώστε όταν αναπτύσσονται καινούριε ε, φυτικές ποικιλίε, ε, οι ασθένειες, ε, η χρήση, η χρήση των υδατινών πόρων, η αντίσταση στις ασθένειες είναι παράγοντες που πρέπει να ελέγχονται. Επίσης πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά για την ανάπτυξη νέων φυτικών ποικιλιών. Επίσης το σύστημα πιστοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτοποίηση και την προστασία του φυτικού υλικού και τη σωστή χρήση του από το γεωργό. Για να έχουμε αποτελεσματική ανάπτυξη νέων φυτικών ποικιλιών δεν αρκεί η πρόσβαση στη βιοπικιλότητα αλλά απαιτείται και η τεχνολογία. Ε, και η μόνη τεχνολογία που ελέγχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η τεχνολογία GM, η γενετική μετάλλαξη και πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να έρθουμε και στο πεδίο της γενετικής μηχανικής. Αναφέρεται το Seed World ε, στην έκθεση Σάλμπαρκ. Είναι μια τράπεζα σπόρων, μια τράπεζα διατήρησης και διαφύλιξης ε, του γενετικού υλικού, των γενετικών πόρων. Σε περίπτωση που καταστραφεί ε, ή αποτύχει κάποια εθνική τράπεζα σπόρων. Εμείς θέλουμε να γίνει παραπομπή ε, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, των ε, Γενετικών Πόρων, στο δίκτυο εθνικών τραπεζών σπόρων. Θεωρώ ότι αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για την πρόσβαση στο υλικό γενετικής αναπαραγωγής. Συχνά ακούγεται ότι η παραγωγή των σπόρων και η ανάπτυξη νέων φυτικών ποικιλιών κυριαρχείται, δεσπόζεται από κάποιες πολυεθνικές. Αυτό ίσως ισχύει παγκόσμια, αλλά σίγουρα όχι στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας από την βιομηχανία σπόρων, το 70% του τζίρου προέρχεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια έρευνα μεταξύ των κρατών μελών και η οποία έδειξε ότι πραγματικά έχουμε μικροεπιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Εξαρτάται για ποιο φυτικό είδος μιλούμε. Αν είναι ε, λαχανικά, ίσως είναι μεγαλύτερες οι εταιρείες. Αλλά στα αγροτικά φυτά πραγματικά έχουμε μικροεπιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στο ε, και στην, στην αμπελουργία επίσης. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ε, εμπορευματοποίηση των απορρογικού φυτικού υλικού προσφέρει ίση πρόσβαση σε κάθε επιχείρηση να θέσει σε κυκλοφορία, να θέσει στο εμπόριο τα προϊόντα της και στην Ευρώπη, όπως είπα, έχουμε πολλές μικροεπιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείες, για παράδειγμα, όπου δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία για την εμπορευματοποίηση των ε, για την εμπορική εκμετάλλευση των σπόρων και υπάρχουν ε, μεγάλες επιχειρήσεις που βασίζονται μόνο στις ικανότητες διαφήμισης και εμπορευματοποίησης. Είναι διαφορετική λοιπόν η κατάσταση στην Ευρώπη. Εν τέλει λοιπόν για τη βιοπικιλότητα, Θέλω να κλείσω επαναλαμβάνοντας ότι στην πρόταση της Επιτροπής για τον απαραγωγικό φυτικό υλικό ε, προτείνονται μια σειρά μέτρων για πιο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις παραδοσιακές ποικιλίε, νέες αντιλήψεις έχουν αναπτυχθεί στην αγορά για να ενθαρρύνεται η παραγωγή οποιοδήποτε φυτικού υλικού και η κυκλοφορία του ε, μέσω μικρών ε, επιχειρήσεων, μικροεπιχειρήσεων. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, το καλύτερο που μπορούμε από αυτήν την άποψη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη Γενική Διεύθυνση Σάνκο. Και τώρα ξαναδίνω το λόγο στην Αντιπρόεδρο Πόλσεν. Παρακαλώ, Μαρίτ. Ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, συναδέρφους μου και θα ήθελα να πω ότι είναι κάπως ε, αστείο ε, να ακούσει κανείς τις διάφορες θέσεις Εννοείται ότι δεν πιστεύω ούτε δευτερόλεπτο ότι μία μεγάλη επιχείρηση αυτομάτως είναι κακή και μία μικρή ε, επιχείρηση αυτομάτως είναι καλή. Ε, η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή. Η διατύπωση που χρησιμοποιείς εδώ πέρα, μεταξύ άλλων, βασίζεται στο γεγονός ότι ε, στον τομέα αυτό η μεγαλύτερη γερμανική επιχείρηση, BASF, μετέφερε εκτός Ευρώπης ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, την έρευνά της ε, για τα φυτά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χάνουμε κάποια πράγματα με τη διατύπωση αυτή. Δεν ήθελα να επιτεθώ στις 5-6 μεγάλες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ανακτήσουμε αυτού του είδους την έρευνα. Να έχουμε να είμαστε πιο ε, ανοιχτοί και αν ε, διαβάσετε την ε, παράγραφο 21 στην έκθεσή μου, λέει σαφώς τι ακριβώς θέλω να επιδιώξω. Μία κοινή ευρωπαϊκή βάση ώστε οι μεγάλες, μικρές και μεσές επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Θα χρειαστούμε όμως νομίζω συντονισμένη κοινή βασική έρευνα ε, της οποίας τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα σε όλων των ειδών της επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών σε προϊόντα στην αγορά. Είναι λοιπόν ε, πολλές ε, οι βασικές λεπτομέρειες και μια από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι να διατηρήσουμε ε, την ε, γενετική ε, βιολογική ποικιλομορφία στην Ευρώπη ταυτόχρονα με την ανάπτυξη νέων τεχνικών. Στις 3 Δεκεμβρίου νομίζω ότι είναι η προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών. Ε, ας συμφωνήσουμε όμως να θέσουμε μια Ας ξεκινήσουμε μία ε, επικοδομητική συζήτηση με κατεύθυνση το μέλλον δεν ε, μιλώ για αποφάσεις, ε, μιλώ για ξεκίνημα της συζήτησης, να διατυπώσουμε έξυπνες ερωτήσεις για να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό είναι αποφασιστικής σημασίας για την ε, προμήθεια τροφίμων στον κόσμο, αλλά και για να έχουμε μια καλή ελπίδα να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή ποικιλομορφία και να έχουμε ε, καλή γεωργία. Ας δούμε λοιπόν αν μπορούμε να συνεχίσουμε ε, να το έχουμε αυτό. Αλλά τελικά θα πρέπει να νομοθετήσουμε όχι σχετικά με την τεχνολογία, αλλά με, την, ε, με τα αποτελέσματα της τεχνολογίας. Και να κλείσω με το εξή. Εάν κάποιο θέλει να επισκευάσει ένα σπίτι, χρειάζεται σφυρί. Ένα σφυρί είναι χρήσιμο, αλλά μπορεί και να σκοτώσει και το γείτονα με το σφυρί αυτό. Με αυτή την ε, ε, σύγκριση ήθελα να κλείσω. Η τεχνολογία ε, δεν είναι το θέμα αυτό καθ' αυτό, αλλά το πώς τη χρησιμοποιούμε. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ Μάριτ Πόλσεν. Μία έκθεση πρωτοβουλίας πάρα πολύ σημαντική πραγματικά. Τώρα, συνάδελφοι, έληξε η συνεδρίαση ε, της Επιτροπής Γεωργίας. Θέλουμε ένα πεντάλεπτο για να συγκεντρωθούμε εδώ οι ε, συντονιστές. Θα συνεχίσουμε στις 3 ε, το απόγευμα.